Nous allons reprendre notre réunion. Nous sortons... Ας συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Μόλις ε, ήρθαμε από μια ανταλλαγή απόψεων για την ακτή του ελεφαντοστού. Ξέρουμε ότι η κατάσταση εκεί είναι δύσκολη. Και νομίζω ότι μπορούμε να ζητήσουμε από τη Γραμματεία να προβλέψει για την ημερήσια διάταξή μας, ε, τη μελλοντική, μια ακρόαση ίσως με τον υπεύθυνο ασφαλείας ε, για την περιοχή της Δυτικής Αφρικής, τον εντεταλμένο της, του ΟΗΕ, τον επιτετραμένο μάλλον του ΟΗΕ, για παράδειγμα, ώστε να σκεφτούμε κι εμείς ποια θα είναι η δική μας τοποθέτηση για τη βοήθεια που προσφέρουμε. Και μήπω πρέπει να προβλέψουμε και κάποιο είδους δράση. Ζητούμε λοιπόν να το προβλέψει η Γραμματεία για τη συνάντηση των συντονιστών σε πρώτη φάση. Συνεχίζουμε τώρα με την ημερήσια διάταξη. Έχουμε την έκθεση του κυρίου Μπέρμαν για τις πολιτικές προκλήσεις και τους δημοσιονομικούς πόρους ώστε να έχουμε μια βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2013. Και πάλι τα κράτη-μέλη ε, πραγματεύονται αυτή τη στιγμή ένα νέο δημοσιονομικό πλαίσιο που θα ορίσει τα όρια για τις νέες διαφορετικές, για τις διαφορετικές μάλλον ευρωπαϊκές πολιτικές, και τα κατόφλια του έως το 2020. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να προβέψει κονδύλια για μια βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2013. Οπότε ετοιμάζει εδώ και κάποιου μήνε το σχετικό ε, έγγραφο και γι' αυτό περιμένει και τη συνεισφορά του Κοινοβουλίου για αυτό το πολύ ζωτική σημασία θέμα. Ο κύριο Σαλβαδόρ Γκαρίγκα είναι ο καθήλυνο αρμόδιο ε, εισηγητή. Και ο κύριος Μπέρμαν ετοιμάζει τη δική μας ενισφορά, από την πλευρά της δικής μας επιτροπής. Θα ψηφίσουμε αύριο την έκθεσή του. Οπότε σε πρώτη φάση θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκαρίγα για να μας ε, περιγράψει τις αδρές γραμμές της εκθεσής του και τις βασικές προκλήσεις που θα έχει να αντιμετωπίσει η Ένωση. Και έπειτα θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπέρμαν και στην Επιτροπή και στους βουλευτές που θέλουν να παρέμβουν. Ο κύριος Γκαρίγκα. Για πέντε περίπου λεπτά. <coughs> Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα που με προσκαλέσατε εδώ. Ευχαριστώ και τα μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης και τον συνάδελφο Βέρμαν και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών που μας βοηθάει πολύ εμάς στην Επιτροπή Ισούρη για να καταλήξουμε στην θέση μας όσον αφορά ιδιαίτερα την αναπτυξιακή πολιτική. Υπενθυμίζω ότι η Επιτροπή μας ε, ΣΟΥΡΕ 1 Φεβρουαρίου θα έχει μια ειδική συνεδρίαση προκειμένου να συζητήσουμε για την εξωτερική πολιτική. Η πολιτική ανάπτυξης αποτελεί μέρος αυτής. Στην Επιτροπή μας μέχρι τώρα έχουμε ασχοληθεί με τα πιο τεχνικά ζητήματα, με τη δομή, με την ευελιξία και με τη διάρκεια του επόμενου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Έχουμε ήδη δύο έγγραφα που έχουν παρουσιαστεί. Το ένα για την ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία και το άλλο για τη στρατηγική 2020 και τις επιπτώσεις της στην, στις δημοσιονομικές προοπτικές, ιδιαίτερα όσον αφορά την δομή και τους στόχους του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου. Για μας η ευρωπαϊκή προσθετή αξία θα αποτελέσει έναν οδηγό για τις επόμενες αποφάσεις που θα ληφθούν όσον αφορά τις δαπάνες. Αποτελεί μια πολύ σημαντική ιδέα, φαντάζομαι και για τα μέλη της δικιάς σας Επιτροπής. Έχουμε κάποια αμφιβολία για το κατά πόσο η στρατηγική 2020 θα πρέπει να αποτελέσει μέρος ή να συμπληρώσει τη δομή δαπανών για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Η στρατηγική 2020 εννοείται ότι είναι μια στρατηγική ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Συγχρόνως όμως υπάρχουν και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δαπάνες, εκτός από την ε, ανάπτυξη, που δεν εντάσσονται πλήρως στη στρατηγική 2020, αλλά που πρέπει να αποτελέσουν μέρος των ε, νέων δημοσιονομικών προοπτικών. Αυτό είναι το δίλημα που αντιμετωπίζουμε στην Επιτροπή μας. Από την άλλη τώρα και σε σχέση με την διάρκεια των επόμενων δημοσιονομικών προοπτικών, μιλάμε για 5 έως 5 συν 5 που είναι η πρόταση Μπαρόσο. Και εκεί κάπου μέσα είναι η 7 ετία. Ή η άλλη εναλλακτική λύση που θα ήταν να μην υπάρξει συμφωνία από το Συμβούλιο για ένα νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οπότε τότε θα έπρεπε να επεκτείνουμε τις τρέχουσες δημοσιονομικές προπτικές. Όλα αυτά είναι σενάρια τα οποία εξετάζουμε στην Επιτροπή μας. Όπως και να έχει το πράγμα πάντως και έχοντας αναλύσει και το άγγραφο του συναδέλφου Μπέρμαν, εγώ ως εισηγητής θα ήθελα να συζητήσω μαζί σας και κυρίως να ζητήσω τη γνώμη σας για μερικά θέματα, κυρία Πρόεδρε. Για παράδειγμα, ποια είναι η γνώμη σας για το πώς μπορούμε όσον αφορά την ανάπτυξη να έχουμε ευρωπαϊκή προστιθάμενη αξία. Πώς, αποφεύγοντας επικαλύψεις, έχοντας καλύτερο συντονισμό μεταξύ διαφόρων υπηρεσιών εξωτερικής δράσης και λοιπόν υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα τη γνώμη σας για αυτά γιατί πιστεύουμε ότι έτσι ε, μπορούμε καλύτερα να δείξουμε ποια είναι η προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Αναπτυξιακής Πολιτικής. Έπειτα πρέπει να δούμε τις κλιματικές αλλαγές, πώς θα τις συμπεριλάβουμε, που και αυτές είναι πολύ σημαντικό θέμα για την Επιτροπή σας. Πώς θα συμπεριληφθούν αυτές στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο. Κάτι άλλο που ο συνάδελφος Μπέρμαν θεωρεί πολύ σημαντικό και έχει συμπεριλάβει είναι τι θα γίνει με τις χώρες μεσαίων εισοδημάτων ε, και εσόδων στο μέλλον. Θα έχουμε μια διαφορετική πολιτική που ξεκινάει από την ανάπτυξη αλλά καταλήγει σε εμπορικές ε, συμφωνίες και άρα διαφορετική ε, χρηματοδότηση από αυτήν που έχουμε μέχρι τώρα. Και κάτι που είναι σημαντικό και για τη δικιά μας Επιτροπή αλλά και για τη δικιά σας είναι το εξής. Ποιο είναι το αναγκαίο ποσό για την αναπτυξιακή πολιτική? Αυτό που δίναμε μέχρι τώρα είναι αρκετό, χρειαζόμαστε περισσότερα. Δεν σας κρύβω ότι σε ένα πλαίσιο δημοσιονομικής λιτότητας που εφαρμόζεται ήδη σε διάφορες χώρες μέλη, είναι δύσκολο να βρούμε τρόπο να αυξήσουμε το ποσό στον προπολογισμό για αυτά τα θέματα. Γι' αυτό θα ήθελα να ακούσω τη δικιά σας γνώμη Μήπως θα έπρεπε να ξαναδούμε τις προτεραιότητες των στόχων που είχε μέχρι τώρα η αναπτυξιακή μας πολιτική. Τέλος, για μας που χρόνια έχουμε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, ξέρετε ότι έχουμε τεόνια προβλήματα της κατηγορίας 4, όπως ονομαζόταν μέχρι τώρα. Θα δούμε στο μέλλον πώς θα την ονομάσουμε εξωτερική πολιτική. Εκεί λοιπόν πάντα είχαμε το πρόβλημα της υποχρηματοδότησης. Και πάντα είχαμε μέσα δημοσιονομικής ευελιξίας για να πετύχουμε τους στόχους μας. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτό το μέσο ευελιξίας. Ποιο πιστεύετε ότι πρέπει να είναι το μέλλον του που μέχρι τώρα κάλυπτε τα κενά της κατηγορίας 4. Τέλος, τέλος, ποια είναι η γνώμη σας για κάτι πολύ σημαντικό που είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Τι θα γίνει με αυτό στο μέλλον. Θα συνεχίσουμε να επιμένουμε να συμπεριλαμβάνεται στον κοινοτικό προπολογισμό ή θα το αφήσουμε έτσι σε κρεμότητα όπως έχει μέχρι τώρα μέχρι να επιτευχθεί πολιτική συμφωνία ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Μου είπατε πέντε λεπτά κυρία Πρόεδρε. Εγώ προσπάθησα να συνοψίσω πολύ σύντομα και τα θέματα που συζητάμε στην Επιτροπή Σούρε και που θα οδηγήσουν σε έκθεση της Επιτροπής αυτής που θα αρχίσουμε να ετοιμάζουμε το Φεβρουάριο. Θα υποβληθούν τροπολογίες και 8 Ιουνίου θα ψηφιστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εννοείται ότι το άλλο θέμα που μας απασχολεί είναι η δικιά σας άποψη, τι έχετε εσείς να πείτε για την αναπτυξιακή μας πολιτική και για το μέλλον της. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπέρμαν έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Υπάρχουν ε, βασικά ερωτήματα που θέτει ο εισηγητή από την Επιτροπή ΣΟΥΡΕ για την στρατηγική 2020 και την αναπτυξιακή μας πολιτική στα πλαίσια του προπολογισμού που δεν είναι βέβαια θέμα αυτής της Επιτροπής. Πρέπει να δούμε επίσης τον ρόλο του αναπτυξιακού προπολογισμού, κλιματικές αλλαγές κλπ. Σε αυτό που έχω ετοιμάσει εγώ επικεντρώνομαι στο ότι ο προπολογισμό για την ανάπτυξη πρέπει να καταπολεμάει την φτώχεια πρώτα απ' όλα. Και πρέπει να βελτιωθούν τα ποσά που δίνονταν για αυτό το σκοπό. Η προθεσμία του 2015 για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων τη χιλιετία εμπίπτει στην περίοδο του προσεχούς πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Και θέλουμε όχι τόσο να μιλήσουμε για περισσότερα χρήματα, αλλά για καλύτερη χρήση των κονδυλίων. Η πρόσθετη αξία, άμα θέλετε, είναι από τη μια μεριά η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και δεν μιλώ για χρήματα, να συντονίσει καλύτερα τα πράγματα μεταξύ των κρατών μελών και να φροντίσει ότι τα κράτη-μέλη καταμερίζουν σωστά τους ρόλους τους για να ξέρουμε ποιος κάνει τι. Η Ευρωπαϊκή θα έπρεπε να έχει συντονιστικό ρόλο που δεν τον έχει ακόμα. Με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι θα εξοικονομούσαμε χρήματα. Χρόνια τώρα ζητάμε καλύτερο συντονισμό και δεν τον έχουμε πετύχει ακόμα. Και ο ΣΑ το ζήτησε. Από πότε, από το 2007. Δυστυχώς δεν έχουμε προχωρήσει, γιατί τα κράτη-μέλη θέλουν συντονισμό, αλλά όχι όταν πρόκειται να συντονιστούν μεταξύ τους. Τώρα, η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται και στα πλαίσια μιας άλλης συζήτηση. Είμαστε 28ος ε, με τομείς όπως είναι η υγεία, υποδομές κλπ. Η βασική συζήτηση όσον αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική θα έπρεπε να γίνεται αλλιώς. Εδώ δεν το εξηγούμε αυτό. Εγώ πιστεύω ότι το καλύτερο θα ήταν να έχουμε μεγάλα προγράμματα από κάποιες χώρες από κοινού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης θα έπρεπε να ασχοληθεί περισσότερο με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την δημοκρατία, τις ανθρώπινες αξίες. Αυτή είναι η δικιά μου υπεποίθηση για την κατηγορία 4 τώρα, όπως την ονόμασε ο Γκαρίγκα, η εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ πιστεύω ότι η Επιτροπή μας ολόκληρη πιστεύει ότι χρειάζονται περισσότερα χρήματα. Με το μέσο συνεργασίας για την ανάπτυξη απαιτούνται δαπάνες οι οποίες δεν εμπίπτουν στο Official Development Aid γιατί δεν τηρούνται τα κριτήρια η ανακούφιση από θεομηνίες, η πρόληψη καταστροφών απαιτεί περισσότερα χρήματα για το μέλλον. Διότι οι καταστροφές που έχουμε διαπιστώσει τον τελευταίο καιρό από τις θεομηνίες κλπ. θα προκύπτουν όλο και πιο συχνά εξαιτία των κλιματικών αλλαγών, για παράδειγμα. Γι' αυτό και λέω ότι χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα έπειτα για τις κλιματικές ε, μεταβολές. Επίσης, χρειάζονται περισσότερα χρήματα, τα οποία δεν μπορούν να έρθουν από την ε, αναπτυξιακή βοήθεια. Δεν πρέπει από τα χρήματα της αναπτυξιακής βοήθειας να φροντίζουμε για αυτά τα πράγματα. Έπειτα χρειάζεται περισσότερη ευελιξία. Κάθε χρόνο πρέπει να βρίσκουμε χρήματα από το μέσο ευελιξίας. Άρα πρέπει να υπάρχουν περισσότερα χρήματα εκεί. Τώρα, όσον αφορά την Αφρική, εδώ έχουμε διάφορα μέσα. Τρία διαφορετικά μέσα, αλλά είμαστε αναποτελεσματικοί μέχρι τώρα όσον αφορά τη διοχέτευση πόρων. Το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο και το Μέσο ε, Συνεργασίας για την Ανάπτυξη θα έπρεπε να διαθέτουν περισσότερα κονδύλια και όχι να μειωθεί το συνολικό ποσό θα ήμουν κατά κάτι τέτοιο. Σημαντικό είναι σε αυτή την έκθεση να πούμε και επίσης ότι η επιδότηση εξαγωγών έχει καταλήξει σε ένα σκάνδαλο. Είναι το ένα τρίτο περίπου τώρα από ό,τι ήταν πριν από 10 χρόνια αποτελεί ένα μέσο σήμερα της πολιτικής γεωργίας, αλλά πρέπει να σταματήσει. Χρειάζεται συζήτηση, όπως λέει και ο Γαρίγκα, για την κατάσταση όσον αφορά τις χώρες μεσαίων ε, εσόδων. Τη βοήθειά μας πρέπει να τη δίνουμε εκεί που είναι πιο αποτελεσματική. Βάσει τη Σούνισετ, για παράδειγμα. Όμως τα θεματικά προγράμματα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία. και να επιτρέπουν την βοήθεια στις χώρες μεσαίων εσόδων για να βοηθηθούν στην ανάπτυξή τους. Δεν πρέπει να εμποδίζουμε αυτή την βοήθεια, όπως συμβαίνει συχνά, γιατί τότε όλες οι ευάλωτες ομάδες κινδυνεύουν και θα βρεθούν σε ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση. 2014 με 2020 θα πρέπει να βρούμε νέες μεθόδους χρηματοδότησης. Μόνο οι επιδοτήσεις δεν φτάνουν. Πρέπει να δούμε τις μικρές επιχειρήσεις, τις οικογένειες, τις πιο ευάλωτες ομάδες. Εκατομμύρια άνθρωποι στις αναπτυσσόμενες χώρες περιμένουν πολλά από τέτοια κονδύλια με revolving funds, με εγγυήσει. Περιμένουν ευκαιρίες για να μπορέσουν να ζουν αξιοπρεπώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι στις αναπτυσσόμενες χώρες. Άρα πρέπει να αναπτύξουμε νέες μεθόδους χρηματοδότησης εμείς εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που έχει παίξει σημαντικό ρόλο αλλά πρέπει να κάνει περισσότερα. και τα δάνεια και οι εγγύησει που δίνει είναι σημαντικές. Να ξέρετε ότι για τη γνωμοδότηση αυτή δεν μιλάω τόσο πολύ για το μέλλον της αναπτυξιακής πολιτικής. Στις τροπολογίες θα είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Τι σημαίνει αϊφόρος, για παράδειγμα. Κάποιες τροπολογίες χρειάστηκε να περιοριστούν ή να αλλάξει η διατύπωση. Αλλά τι να κάνουμε, είμαι δημοσιογράφος καταρχήν. Πιστεύω πάντως ότι βοηθάνε οι τροπολογίες. Αυτά, ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα, λέει η Πρόεδρος. Ο Σφανίτε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Να θυμίσω καταρχήν ότι η Κομισιόν ήδη έδωσε γραπτός απαντήσεις την προηγούμενη φορά επί του σχεδίου νομοδότησης όπου χαιρετίζει η Κομισιόν εν πωλής τις ε, προτάσεις του εισηγητή. Ειδικότερα συμφωνούμε με τα αιτήματα και τις ιδέες που αφορούν το, την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας και την ε, συνέχιση του Ταμείου Ανάπτυξης ακόμα και αν εγγραφεί στον προϋπολογισμό, ε, το μέσο ευελιξίας για κρίσεις, το στόχο ενίσχυσης της πολιτικής για ανάπτυξη στα πλαίσια της νέας συνθήκης, την ανάγκη διαφοροποίησης αλλαγή της φύσης των εταίρων, παίζει ρόλο εδώ, και όπως είπα, διερεύνηση καινοτόμου χρηματοδότησης όπως συνένωση, ομαδοποίηση πόρων και επιχορηγήσεων και η Κομισιόν ενδιαφέρεται επίσης στην περαιτέρω εξέλιξη του ρόλου του δωρητή για το συντονισμό των κρατών μελών. Ε, τώρα, πιο συγκεκριμένα για τώρα, δεχόμεθα τα γεωγραφικά όρια που πρέπει να ξεπεραστούν για τους ε, χρηματοδοτικούς μηχανισμούς. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δούμε πιο συνεκτικά την Αφρική και στηρίζομαι και την ε, ατζέντα υπηρετικής ολοκλήρωσης. Πιστεύω όμως ότι η καλά εδρεωμένη πολιτική γειτονία δικαιολογεί και συμπληρώνει και εφαρμόζει και μελλοντικές πολιτικές στο μέλλον με πιο διασυνδεδεμένα μέσα ή μηχανισμούς όπως το MPI, το DCI, το μηχανισμό για την ε, αναπτυξιακή συνεργασία κλπ. Θέλουμε βέβαια τις δαπάνες, ε, θέλουμε οι δαπάνες ε, να έχουν στόχο την ανάπτυξη οικονομική και κοινωνική των παραληπτών. Επίσης ε, θέλουμε ε, να ε, βελτιωθούν οι γραμμές του προϋπολογισμού για την αναπτυξιακή βοήθεια. Είναι σημαντικό αυτό γιατί επηρεάζονται οι εταίροι μας και στις αναδυόμενες οικονομίες. Είναι όλο και πιο σημαντικό να υποστηρίξουμε τις πολιτικές της Ένωσης στη σφαιρική τους διάσταση και αυτό χρειάζεται ευελιξία ε, σε σχέση με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων. Επίσης θέλουμε συλλογική δέσμευση για να επιτευχθεί το 7% ε, του καθάριστου εθνικού προϊόντος ε, για την ανάπτυξη με στόχο τις πιο ευάλωτες. Να πω και δύο λόγια για μία από τις τροπολογίες που προτείνονται, η τροπολογία 20 που ζητάει χωρίς τη, χωριστό ε, κεφάλαιο για θέματα κλίματος. Εμείς θέλουμε να είναι πρόσθετα τα ταμεία και η χρηματοδότηση για το κλίμα. Η Κομισιόν εξετάζει το θέμα της κλιματικής αλλαγής, το οριζόντιο θέμα, τουλάχιστον στην οικογένεια Ρέλεξ, είναι ότι τα οριζόντια θέματα που αφορούν τις χώρες εταίρους θα πρέπει να ενταχθούν στην εξωτερική δράση με γεωγραφική βάση και από την άλλη πλευρά αληθεύει ότι η κλιματική αλλαγή είναι ένα ε, κύριο ε, γενικό θέμα και πρέπει να το δούμε χωριστά Πράγμα που μπορεί να μας κάνει να σκεφτούμε μήπως χρειάζεται ένα χωριστό, ένα, να χρειάζεται ένας χωριστός μηχανισμός. Πιστεύουμε ότι αυτό θα πρέπει να είναι στον τίτλο εξωτερική ε, βοήθειας, ούτω ώστε να συντονίζονται οι δράσεις μας στις χώρες εταίρους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκέρινς έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι η πρώτη φορά που μας δίνεται ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Θα είμαι σύντομος. Θα περιοριστώ σε μερικές μόνο παρατηρήσεις. Ευχαριστώ και τον Τέις και τον κύριο Καρίγα που μας εισήγαγαν στη συζήτηση. Με μεγάλο ταλέντο. Μας διευκολύνει τη ζωή αυτό γιατί έθεσαν τα ζητήματα πολύ ξεκάθαρα τι προστιθέμενη αξία μπορούμε να περιμένουμε από την ε, πολιτική συνεργασία για την ανάπτυξη. Πολύ βασικό ερώτημα. Αλλά πρέπει να απαντήσουμε με νούμερα. Οι συνέπειες μακροοικονομικά της αναπτυξιακής μας πολιτικής μπορεί να μετρηθεί βάσει της προστιθέμενης ανάπτυξης οι συνέπειες της δράσης δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις υπονάπτυξη χώρες. Από την άλλη μεριά μπορούμε να κάνουμε τον απολογισμό τι έχει γίνει με τις εκστρατείες εμβολιασμού, τι έχει γίνει με ανθρωπιστική βοήθεια και να δούμε έτσι ποια είναι τα αποτελέσματά μας. Αξιολογήσεις γίνονται και δείχνουν τα βασικά στοιχεία. Για σύντομα, το 2020 θα μπορούμε να πούμε τι πετύχαμε με την πολιτική μας το 2010. Γιατί αυτά τα οποία θέλετε να πετύχετε το 2015, ε, ξεκινάτε ένα έργο με ένα νοσοκομείο και βλέπετε ότι έχει ξεκινήσει να δουλεύει. Αλλά δεν μπορούμε εκ των προτέρων να πούμε και ούτε και την ίδια στιγμή μπορούμε να πούμε κατά πόσο αποφέρει καρπού η πολιτική μα. Είναι πολύ αργότερα που το ξέρουμε αυτό. Αλλά έπειτα υπάρχει και ένα άλλο τρόπο που δεν ε, έχει ποσοτική έκφραση νούμερα. Αποφεύγουμε ένα πόλεμο. Πώ θα το υπολογίσει αυτό με οικονομικού όρου, Δεν μπορεί να το μετρήσει, δεν μπορεί να μιλήσει με ποσά. Τι κέρδισε από την αποφυγή. Ένα χρόνο ειρήνη. Πόσο στοιχίζει. 50 εκατομμύρια γυναίκες που βρήκαν λίγη αξιοπρέπεια. Αυτό πόσο κοστίζει. Πάρα πολύ. Αλλά ποσοτικά δεν μπορούμε να το εκφράσουμε. Άρα πρέπει να δούμε διαφορετικά τον τρόπο με τον οποίο κρίνουμε αυτά που πετύχουμε. Γιατί τα νούμερα, η ποσοτική έκφραση είναι μόνο ένα μέρος της αξιολόγησης που κάνουμε. η απελευθέρωση ενός λαού, μιας κοινότητας, ενός χώρου, μια κυβέρνηση που βρίσκει τη θέση της ενώ δεν υπήρχε πια. Είναι πολύ περίπλοκα τα πράγματα. Το είδαμε και στην ακτή ελεφαντοστού. Εννοείται. Πώς να μετρήσεις την ανάπτυξη αυτή. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθήσαμε και αυτή είναι η προστιθέμενη αξία της δικιάς μας βοήθειας. Να έχουμε δηλαδή μια όλο και πιο στενή συνεργασία και σχέση με την ε, περιοχή βασιζόμενη ε, στο Ταμείο Ανάπτυξης. Όμως, θέλω να ζητήσω να έχουμε μια επιστημονική βάση γιατί αυτό μας λείπει. Το είπα και τις προάλλες. Η Γενική Διεύθυνση Συνεργασία και Ανάπτυξη συγχωνεύτηκε. Δημιουργήθηκε ένα κενό το οποίο όμως δεν καλύφθηκε. Χρειαζόμαστε έναν πυρήνα ερευνών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε επιστημονικά να λαμβάνονται οι αποφάσεις οι οποίες θα καταλήγουν στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλιώς, όπως συνέβαινε και κατά το παρελθόν, έτσι και τώρα θα ακούμε τι λένε οι άλλοι. Που μπορεί να έχουμε κάθε σεβασμό σε αυτούς, ε, παγκόσμια τράπεζα κλπ. Όπως έγινε και με τις αγροτικές τιμές η Παγκόσμια Τράπεζα τι επέβαλε. Και εμεί δεν έχουμε να αντιπαραθέσουμε τίποτα, άρα δεν έχουμε παρά να δεχτούμε ό,τι λένε αυτοί. Αφού δεν έχουμε τίποτα να προτείνουμε εμεί. Τέλος, ΦΕΔ και πώς συμπεριλαμβάνεται στον προπολογισμό. Σας έχω εξηγήσει ότι δεν συμφωνώ με το πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνεται αυτή η συζήτηση. Αν γίνει αυτό, συμφωνώ μόνο εφόσον δεν θα έχουμε τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που περιμένουμε. Γιατί μπορεί να γίνει με τέτοιο τρόπο που να είμαστε αντιπαραγωγικοί. Ξέρουμε ότι δίνουν 27 χώρες για την τροφοδότηση του Αναπτυξιακού Ταμείου. Οπότε είναι η οροφή συν χ. Κάποιοι εκπρόσωποι από τα κράτη-μέλη μου λένε ότι αν το Ευρωπαϊκό Ταμείο ανάπτυξη μπει στον προπολογισμό, τότε θα μειωθούν αντίστοιχα οι συνεισφορές των χωρών μελών που είναι στάξος του 1.02. Οπότε τότε θα είναι οροφή μείον χ. Πράγμα το οποίο θα μας οδηγούσε να βάλουμε σε αντιπαράθεση την αναπτυξιακή πολιτική με όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό εγώ δεν θέλω να μιλάμε για ψηλοοικονομίες ενώ Συμβούλιο Υπουργών Ανάπτυξης δεν υπάρχει. Καλά καλά. Να δούμε λοιπόν καλύτερα σε τι πλαίσιο φτιάχνουμε την ε, πολιτική συνεργασία και για την ανάπτυξη και να δούμε πώς αυτή λειτουργεί. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ξέρει ότι το πλαίσιο και συγκυρία δεν είναι τόσο θετική για να γίνει για να συμπεριληφθεί ακριβώς στον προπολογισμό το ΦΕΔ κάθε Εθνικό Κοινοβούλιο έθεσε κοινοβουλευτική ερώτηση στον Υπουργό του Οικονομικών για να δούνε εφόσον συμβεί αυτό ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην τροφοδότηση του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού. Δεν ξέρω τι είπαν, αλλά μπορώ να φανταστώ. Αν γίνει λοιπόν αυτό, θα δημιουργηθούν περισσότερα προβλήματα από ό,τι θα λυθούν. Καήκαμε δηλαδή. Και τέλος, εφόσον συμπεριληφθεί στον προπολογισμό το ΦΕΤ, τότε θα εξαφανιστεί και μια μορφή συναπόφασης ανάμεσα στους Αφρικανούς και τους Ευρωπαίους. Η... Τι θα γίνει λοιπόν με αυτήν ε, τη συνήθεια που έχουμε να έχουμε διάλογο για το DCI. Το μέσο συνεργασίας για ανάπτυξη. Δεν θα μπορούσαμε να δώσουμε χρήματα για τις peace facilities στην Αφρική που μας επέτρεψαν να παίξουμε σταθεροποιητικό ρόλο στην περιοχή του Ταφούρ. Εδώ, και μιλάω εδώ για ένα πρόβλημα που μου δημιούργησε πολλές ανησυχίες παλιότερα. Δεν ήμουν σίγουρος. Τώρα πιστεύω ότι είναι κάτι θετικό. Αν έχουμε και τη συμφωνία από τις χώρες ΑΚΕ, είναι προτιμότερο, γιατί έτσι νιώθουμε ότι είναι μια απόφαση που στέκει. Που βασίζεται σε ένα πνεύμα συνεργασίας. Αλλιώς να μην μιλάμε για προστιθέμενη αξία, αν δημιουργούμε προβλήματα εκεί που προς το παρόν δεν υπάρχουν. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη. Λίγα σχόλια θα κάνω μόνο για την έκθεση του κυρίου Μπέρμαν. Συμφωνώ σε γενικές γραμμές, υπογραμμίζω όμως δύο θετικότατα σημεία. Το ένα είναι η πρότασή του για ενιαίο χρηματοδοτικό μέσο για την Αφρική. Άρα θα είναι πιο εύκολο να εφαρμοστούν οι πολιτικές μας και συμμερίζομαι στην αυστηρή κριτική που κάνει στις εξαγωγικές επιδοτήσεις. Όμως, επιτρέψτε μου κάποια σημεία να θέλω να τα προχωρήσουμε και να τα επεξεργαστούμε περισσότερο. Μιλάτε για περισσότερη και καλύτερη βοήθεια. Νομίζω ότι πρέπει να δεχτούμε ότι πολλά κράτη-μέλη δεν καταφέρνουν να ανταποκριθούν στις υφιστάμενες δεσμεύσεις τους. Πιστεύω επίσης ότι τώρα υπάρχει ανάγκη να αναπτύξουμε κάποια καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα και μηχανισμούς. Όχι ε, υποκαθιστώντα άλλα. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο θέμα φόρων. Υπάρχουν τομεί που ωφελούνται από την παγκόσμια οικονομία και αυτοί οι τομείς ε, αναλαμβάνουν κοινωνικές ευθύνες ε, για οικονομική και κοινωνική σταθερότητα. Θα ήθελα λοιπόν να μπει το θέμα του φόρου των οικονομικών συναλλαγών, χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Ε, είναι σημαντικό αυτό για να αντιμετωπίσουμε καινοτόμα τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς. Μιλάτε για καλύτερη βοήθεια. Και εδώ νομίζω ότι μπορούμε να επεξεργαστούμε περισσότερο την έκθεσή σας. Ένας λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε να ε, εκπληρώσουμε τους στόχους της χιλιετίας είναι, και πρέπει να το δεχτούμε αυτό, δεν ε, αναγνωρίζουμε το περιβάλλον, τους φυσικούς πόρους, τα οικοσυστήματα και τη συμβολή τους ε, στην ανάπτυξη του ανθρώπου και στην εξάλληψη της φτώχειας. Τώρα, αν είναι σωστά τα στοιχεία μου, μόνο 3% της επίσημης βοήθειας πάει σε περιβαλλοντικά θέματα. Τα περιβαλλοντικά θέματα θα πρέπει να είναι ορατά και να αποτελούν τμήμα των εξωτερικών πολιτικών και των χρηματοδοτικών μηχανισμών μέσων. Θέλω λοιπόν να επικεντρώσω τα συμπεράσματά μου σε δύο σημεία. Πρέπει να πούμε σαφέστερα ότι η βοήθεια δεν εστιάζει ε, σαφώς στην εξάλληψη της φτώχειας και την αηφόρο ανάπτυξη. Και ένα τελευταίο σημείο που δεν μπορούμε να αποφύγουμε είναι ότι η καλύτερη βοήθεια συνεπάγεται κατά πολέμηση των φορολογικών παραδείσεων που οδηγούν σε φοροαποφυγή, διαφυγή και διαφυγή κεφαλαίων από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, στηρίζω απόλυτα την έκθεση του συναδέρφου Τάις Μπέρμαν. Εννοείται ότι μπορεί να εμπλουτιστεί με σχόλια, όπως αυτά της κυρίας Γκρέης. Κάποια από τα σημεία που ανέφερε η συνάδελφος, νομίζω ότι είναι σημαντικά και απόλυτα συνεκτικά με την έκθεση του ΤΑΙΣ. Όλα όσα έχουν να κάνουν με τους νέους μηχανισμούς, δηλαδή εσόδων. Όλα αυτά αντιστοιχούν απόλυτα στην ε, δικιά μας φιλοσοφία και του εισηγητή. Έχω να κάνω τρία-τέσσερα σχόλια. Πρώτον, θέλω να αντιδράσω στις ερωτήσεις του συναδέλφου Γαρίγα. Όταν έθεσε το θέμα της προστιθέμενης αξίας, δεν μιλούσε ακριβώς για το έτσι όπως αντέδρασε ο Γκέρενς. Δηλαδή η αναπτυξιακή βοήθεια, τι προστιθέμενη αξία προσφέρει. Νομίζω ότι αυτό που ρώτησε ο Σαλβαδόρ Γαρίγα είναι ποια είναι η προστιθέμενη αξία από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναπτυξιακή βοήθεια σε σχέση με τις συνέπειες που έχει η αναπτυξιακή βοήθεια από την κάθε μας χώρα χωριστά. Ότι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιο αποτελεσματική, πιο παραγωγική όσον αφορά την ανθρωπιστική της βοήθεια από ότι η αντίστοιχη βοήθεια χωριστά της Ισπανίας, ε, της Γαλλίας και ξέρω εγώ τι. Η προστιθέμενη αξία, η πιο σημαντική, είναι ο εξευρωπαϊσμός της συνεργασίας ανάπτυξης. Γιατί έτσι υπάρχουν χώρες οι οποίες εξορισμού, πέρα από το ότι μερικές είναι πιο γενναιόδερες, με την ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια όλες μαζί οι χώρες μας βοηθάνε περισσότερο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη συνεργασία της για την ανάπτυξη μπορεί επίσης να βάλει κάποιες προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ οι επιμέρους χώρες στις συμφωνίες συνεργασίας δεν το κάνουν. Γιατί τότε τίθεται πολλές φορές θέμα γνωριμιών, καλών φίλων, εκατέρωθεν κλπ. Για να είναι μέγιστη η προσθεθέμενη αυτή αξία, πρέπει να χρησιμοποιούμε την υπηρεσία εξωτερικής δράσης όσο γίνεται καλύτερα. Μην ξεχνάμε ότι η μεγαλύτερη εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εξωτερικό είναι σε υποανάπτυξη χώρες. Είναι εκεί δηλαδή όπου η συνεργασία μας βασίζεται σε προγράμματα υπέρ της ανάπτυξης. Δεύτερο σχόλιο. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον άκουσα τον προβληματισμό του κύριου Γαρίγα για τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε σε χώρες μεσαίων εσόδων. Είναι ένα πρόβλημα. Πολύ περισσότερο όμως πρέπει να προβληματιστούμε για την αναπτυξιακή βοήθεια και την συνεργασία μας σε χώρες του Νότου αναδυόμενες με τεράστιες δυνατότητες εξέλιξης. Αλλά όπου πλήττω από τεράστιες ανισότητες στο εσωτερικό τους. Δεν θέλω να αναφέρω συγκεκριμένα χώρες, να κατονομάσω χώρες, μην έρθει μεθαύριο πρέσβης και με κολλήσει στον τοίχο, αλλά είναι αλήθεια ότι έχω παράδοση. Ξέρω από μη κυβερνητικές οργανώσεις της Ισπανίας και της Πορτογαλίας ότι έχουν παράδοση να δρούν σε κάποιες χώρες της Λατινικής Αμερικής ως υπερδυνάμεις. Και δρούν προσπαθώντας να απαλείψουν την ένδια, ενώ η προτερότητα δεν μπορεί να είναι η παρέμβαση απ' έξω, όταν υπάρχει δυνατότητα σε εσωτερικό ή περιφερειακό επίπεδο. Γι' αυτό να αναπτύσσουμε μηχανισμούς συνεργασίας που να αντικαταστούν την ε, γενική ε, πολιτική παρέμβαση ανάπτυξης με ε, παρέμβαση για την ανάπτυξη σε διάφορους τομούς συγκεκριμένα. Τρίτο σχόλιο. Άκουσα τον Σαλβαδόρ Γαρίγα με πολύ ενδιαφέρον να αναφέρεται στα διάφορα σενάρια των δημοσιονομικών προπτικών. Εγώ δεν ήξερα ότι συζητούσαμε μόνο το 5 και το 5 συν 5 και το 7, αλλά ακόμα ότι υπάρχει και το σενάριο του να μην υπάρχει χρονικός προσδιαρισμός και να προχωράμε χρόνο το χρόνο. Θέλω να μου επιβεβαιώσει, έτσι είναι. Καλά το κατάλαβα. το Ταμείο Ανάπτυξη τώρα. Σωστά τα λέει ο κύριο Γκέρι, αλλά το πιο ανησυχητικό είναι ότι οι χώρε με τι οποίε δουλεύουμε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξη δεν θέλουμε να συμπεριληφθεί στον ε, κανονικό προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί πιστεύουν ότι τότε θα μειωθούν τα κονδύλια στα οποία βασίζονται. Ολοκληρώνω κυρία Πρόεδρε. Πιστεύω ότι έχει επιτευχθεί μεγάλη πρόοδος. Οι συνάδελφοί μας που εργάζονται στον προϋπολογισμό έχουν κερδίσει την ε, εμπιστοσύνη μας. Πριν από 12 χρόνια περίπου δεν ήταν έτσι. Και δεν υπήρχε και το κύρος αυτό παλιά στην ε, συνεργασία για την ανάπτυξη. Η πολιτική αυτή ήταν λιγάκι ελεημοσύνη, ανθρωπιστική βοήθεια. Τώρα έχει αποκτήσει ιδιαίτερο κύρος. Παλιά δεν θεωρώταν θέμα προτεραιότητας. Τώρα είναι, έχει αρκετή προτεραιότητα, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρχει συνέχεια. Ευχαριστώ λοιπόν τον Σαλβαδόρ, γιατί οι συνάδελφοι, σαν και αυτόν, έχουν βοηθήσει πολύ να επιτευχθεί αυτό το πνεύμα. Και το τελευταίο, off the record, κυρία Πρόεδρε. Κάποιοι, κάποιος ξέχασε τα γυαλιά του εδώ. Οπότε να περάσει να τα πάρει. Είναι γυαλιά μια γνωστής μάρκας και αυτός που τα άφησε προφανώς δεν βλέπει τώρα. Δεν ξέρω τι διαδικασία υπάρχει για να επιστρέφονται, να επιστρέφουμε την όραση σε κάποιον που την έχει χάσει. Δεν ξέρω, μπορεί η γραμματεία να ξέρει ποιον είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ το λέω να το ξέρει η γραμματεία ότι τα γυαλιά κάποιου βρίσκονται εδώ. Κάποιο έχει ξεχάσει εδώ τα γυαλιά Ο κύριο Κόρτη Γάστρα έχει τώρα το λόγο, λέει πρόεδρο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Και εγώ συγχαίρω τον εισηγητή μας τον κύριο Πέρμαν για την εξαίρετη γνωμοδότησή του. Ευχαριστώ πολύ και τον Σαλβαδόρ Γαρίγα. Η δουλειά που κάνει στην Επιτροπή Σούρε είναι πάρα πολύ σημαντική. Συγχαίρω τον εισηγητή μας πάνω απ' όλα γιατί υπογραμμίζει στην έκθεσή του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τηρεί τις δεσμεύσεις της και τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την πολιτική ανάπτυξης. Αυτό λέγεται και στην Λισαβόνα και πρέπει να το επενθυμίσουμε. Οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως δυστυχώς είναι περιορισμένοι, κυρίως σε θέματα ανάπτυξης. Και θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι αν επικεντρωθούμε στις χώρες χαμηλότερων εισόδων, θα κάναμε καλά. Αλλά μην ξεχνάμε τους πιο φτωχούς πληθυσμών άλλων χωρών στη Λατινική Αμερική. Συνεπώς, Σαλβαδόρ, η δουλειά σου είναι πολύ καλή. Δεν είναι εύκολο να στηρίξει κανείς τις αναπτυξιακές πολιτικές στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως έχουμε αναλάβει κάποιες υποχρώσεις και θέλουμε να μείνουμε σε αυτές. Και εμείς, οι Ευρωπαίοι πολίτες, αλλά και οι πολίτες των χώρων που υποφελούνται από τη βοήθεια αυτή δεν θα καταλάβουν αν αλλάξουμε κάτι. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα να πετύχουμε το 0,7% να είναι το ποσοστό για την αναπτυξιακή βοήθεια και θα ήθελα να φαίνεται αυτό στο τελικό κείμενο της έκθεσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Κύριε Κέλλερ τώρα. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι μια σαφέστατη προστιθέμενη αξία της αναπτυξιακής πολιτικής, δυνητικά έστω, είναι το θέμα του συντονισμού. Δεν υπάρχει άλλο επίπεδο στον κόσμο που να λειτουργεί τόσο καλά ε, ο συντονισμός όσο σε επίπεδο ένωσης. Πρέπει να βελτιωθούμε εδώ. Τώρα για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια και την ευελιξία. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να φροντίσουμε η επίσημη βοήθεια, η αναπτυξιακή βοήθεια, να εντάσσεται σε αναπτυξιακά έργα που θα λειτουργούν με τα σωστά κριτήρια. Τώρα έχουμε αυτό το 10% κόστος δηλαδή που μπορεί να είναι κάτι άλλο από επίσημη βοήθεια, εκτός από επίσημη βοήθεια. Και θέλω μια καταγραφή του τι είναι το 10% και τι είναι το 90%. Γιατί καμιά φορά Μπερδεύονται τα κριτήρια είναι στο 90% ή στο 10%. Πόσο πολύ είναι αυτό το 10%, τι καλύπτει. Καλό είναι λοιπόν κάποια στιγμή να γίνει αυτή η δουλειά. Επίσης, η ευελιξία που τη συζητάμε πολύ μπορεί να πάει και προς την άλλη κατεύθυνση. Γιατί να μην πάρουμε κάτι που δεν έχει χρησιμοποιηθεί στη γεωργία και να το πάμε στην ανάπτυξη ή και το αντίστροφο. Γιατί να γίνεται μόνο το αντίστροφο. Στην Επιτροπή ΝΤΕΒΕ δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο το αναπτυξιακό κομμάτι των δημοσιονομικών προοπτικών, να βλέπουμε και άλλα τμήματα, όπως είπε και ο κύριος ε, Μπέρμαν, ε, εξαγωγικές επιδοτήσεις και άλλες επιδοτήσεις στο γεωργικό τομέα. Πού πάνε τα λεφτά, σε άλλους τομείς. Να το βλέπουμε αυτό γιατί οι περισσότεροι από αυτούς τους τομείς έχουν εξωτερικές διαστάσεις που δεν έχουμε δει. Αυτό πρέπει να το κάνουμε. Όχι μόνο να βλέπουμε την πολιτική, τους τομείς της πολιτικής, αλλά και τον προϋπολογισμό. Αυτό είναι δύσκολη δουλειά, αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε. Και για τα χρηματοδοτικά μέσα και μηχανισμούς ε, που τώρα γίνονται διαβουλέσεις πάνω σε αυτά στην Κομισιόν πρέπει να συμμετέχουμε. Ε, διάμεση αξιολόγηση της DCI του χρηματοδοτικού μέσου για την αναπτυξιακή συνεργασία και, και αλλού όταν υπησέρχονται θέματα προϋπολογισμού όχι μόνο για την ανάπτυξη αλλά και σε άλλα κεφάλαια, σε άλλους τομείς. Ο κύριος Φένσον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν από λίγο καιρό κάναμε μία ακρόαση για το θέμα αυτό στην ε, Βόρεια Αφρική. Και ακούσαμε ότι υπήρχαν κάποιοι ενδιασμοί για τους αριθμούς που παρατέθηκαν, τα αριθμητικά στοιχεία, και ιδίως ό,τι αφορά τις θέσεις εργασίας που χρειάζεται Ξέρουμε ότι το ίδιο ισχύει και στι περιοχέ νοτίω τη Σαχάρα τι τελευταίε εβδομάδε. είδαμε σε τι απελπισία έχουν περιέλθει οι νέοι. Λόγω χάρη, α θυμηθούμε την Τινησία. Θεωρούν ότι δεν έχουν μέλλον, ζουν πραγματικά σε απελπισία. Πιστεύω λοιπόν, Πρόεδρε, ότι θα πρέπει εδώ να τολμήσουμε να τολμήσουμε να μιλήσουμε με τους επιχειρηματίες, να μιλήσουμε με τους εργοδότες και να επενδύσουν στις χώρες τους. Είναι προφανής προτεραιότητα αυτή για μας. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης για τις νέες γενιές των αναπτυσσόμενων χωρών. Θα πρέπει λοιπόν να προσελκύσουμε περισσότερους από έναν εργοδότη, έναν επενδυτή που έχουμε κάνει ως τώρα. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Και τώρα περνάμε στην τελευταία φάση εξέταση του θέματο. Έχουμε καθυστερήσει λίγο. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκαρίγα και στον κύριο Μπέρμαν για τρία-τέσσερα λεπτά περίπου κατά τον καθένα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το συμπέρασμά μου είναι ότι σημειώνω τις ανησυχίες των συναδέλφων. Θα αναφερθώ όμως συγκεκριμένα σε τρία σημεία που μου φάνηκαν πολύ ενδιαφέροντα για την έκθεση. Πρώτον, η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία των πολιτικών συνεργασίας για την ανάπτυξη. Όπως λένε και οι συνάδελφοι, από τη μια είναι σημαντικό να το δούμε αυτό σαν ένα γενικό μέσο αξιολόγησης για να δούμε πόσο σημαντική είναι η αναπτυξιακή πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαντάζομαι ότι εκφράζεται ποσοτικά, εσείς είσαστε πιο ειδικοί από μένα στην αναπτυξιακή πολιτική, εγώ είμαι ειδικό στον προπολογισμό, αλλά ό,τι μπορεί να βελτιώσει μια κυβέρνηση, μια δίκηση, να μειώσει την φτώχεια, να βοηθήσει κοντινές ή μακρινές χώρες, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία έχουν αντίκτυπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους πολίτες της, οπότε δεν χρειάζεται να βρούμε άλλους τρόπους και άλλες κοινοτικές πολιτικές. Συγχρόνως όμως έχει δίκιο ο Μιχελ Άγχελ για το ότι για να εκφραστεί ποσοτικά η προστιθέμενη αυτή αξία είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε κατά πόσο η αναπτυξιακή πολιτική θα χρηματοδοτείται από 27 διαφορετικούς εθνικούς προπολογισμού ή θα πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας κοινή αναπτυξιακής πολιτικής των ε, χωρών μελών και κατά πόσο η δεύτερη αυτή περίπτωση είναι περισσότερο αποτελεσματική. Αυτό το έχουμε κάνει στην πολιτική έρευνας και εκεί είναι ξεκάθαρο ότι αν χρησιμοποιηθούν χρήματα από έναν κοινοτικό προϋπολογισμό ενιαίο, αυτό είναι πολύ προτιμότερο, έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα από ότι αν η κάθε χώρα δίνει ξεχωριστά. Πολλοί αναρωτήθηκαν αν το ίδιο ισχύει και στην αναπτυξιακή πολιτική. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα επειδή περνάμε καιρούς λιτότητας. που θα ισχύουν και στις διαπραγματεύσεις των επόμενων δημοσιονομικών προοπτικών. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η προστιθέμενη αξία μιας κοινή αναπτυξιακής πολιτικής. Γιατί θα αποτελέσει διαπραγματευτικό χαρτί για μας, όπως καταλαβαίνετε με τα κράτη-μέλη, για να αποφασίσουμε για τα τελικά ποσά που θα έχουν προορισμό την αναπτυξιακή βοήθεια. Κάτι άλλο για τον κύριο Μαρτίνες. Με ρωτήσατε για τα σενάρια που κυκλοφορούν όσον αφορά τη διάρκεια των επόμενων δημοσιονομικών προπτικών. Υπάρχει και το σενάριο της μη απόφασης για χρονική διάκρια, διάρκεια. Ξακολουθεί να εφίσταται ως πιθανότητα αυτό το σενάριο. Ακούγεται από πολλές πλευρές. Ως εισηγητή Τη πάντω για τι δημοσιονομικέ προοπτικές σα λέω ότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε κοινοτικό προπολογισμό με λιγότερα ποσά από αυτά που έχουμε τώρα. Όσο κι αν εξοικονομήσουμε, είναι δύνατον να έχουμε μια πολιτική έρευνας, μια πολιτική συνοχής, μια γεωργική πολιτική ή μια πολιτική ανάπτυξης με χαμηλότερα ποσά. Αυτό το λέμε. Και δεν μπορεί να γίνεται ετήσια διαπραγμάτευση. Και δεν είναι αυτό που θα γίνει αν δεν υπάρξει απόφαση. Είπαμε ότι θα παρατείνουμε την τωρινή κατάσταση τον επόμενο χρόνο ή το μεθεπόμενο όσο δεν υπάρχει συμφωνία πολιτική. είπαμε ότι μεγαλύτερες πιθανότητες κλείνουν προς τα 5 χρόνια, τα 5 συν 5 ή τα 7. Από τις αντιδράσεις των συναδέρφων πάντως, καταλαβαίνω ότι περισσότεροι θέλουν το status quo. Ότι αυτό είναι προτιμότερο για το μέλλον. Αυτά είναι τα συμπεράσματα που είχα να αναφέρω, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπέρμαν τώρα. Κυρία Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά την προστεθεμένη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αναπτυξιακή της πολιτική, έχω την εντύπωση ότι πρέπει να έχουμε πάντοτε υπόψη τους, τρίτους, τους τρεις στόχους που θέτουμε πάντοτε στην διεθνή πολιτική, τουλάχιστον κατά τη δική μου άποψη. Πρέπει να σκεπτόμαστε για τα παιδιά μας και τα παιδιά των άλλων να εξασφαλίσουμε την ειρήνη. Μια παγκόσμια τάξη που να είναι βασισμένη στα δικαιώματα για όλους τους πολίτες και χρειάζεται να γίνουν όλα αυτά σε έναν κόσμο που θα προστατεύουμε το περιβάλλον και θα διαφυλάσσουμε τους πόρους μας. Είναι τρεις απαιτήσει αυτές. Η ειρήνη, το δίκαιο και ε, το περιβάλλον. Ε, είναι ε, αδύνατο μια χώρα να το πετύχει αυτό μόνη της. Είναι αδύνατο να το πετύχει χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την ειρήνη πρέπει να συνεργαστούμε στενά παγκοσμίως. Για τα δικαιώματα των πολιτών η Ευρωπαϊκή Ένωση που δεσμεύεται να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν περισσότερο την ισότητα για όλους η Ευρωπαϊκή Ένωση που ακολουθεί τις δικές της αρχές, τις δικές της αντιλήψεις, μπορεί να έχει τέτοιες προσδοκίες, αλλά με το 7% του παγκόσμιου πληθυσμού και το 7% της ε, παγκόσμιας οικονομίας μπορούμε κάτι να καταφέρουμε εάν συνεργαστούμε. Και το ίδιο για το περιβάλλον. Εδώ ο προπολογισμό της ανάπτυξης είναι καθοριστική σημασίας ως εργαλείο προκειμένου να παρέμβουμε στις χώρες που είναι πολύ φτωχές, που δεν μπορούν να τα καταφέρουν μόνοι τους προς στιγμή. Τα κράτη-μέλη, όπως είπε η Κατρίν πολύ σωστά, τα κράτη-μέλη οφείλουν να κάνουν όσα υποσχέθηκαν. Ιδάλλως, εάν δεν καταβάλουν το 0,7% του ΑΕΠ τους, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδείξει ότι με το δικό τη τον προπολογισμό, με ένα ενιαίο εργαλείο μπορεί να κάνει τη διαφορά σε αυτέ τι αναπτυσσόμενε χώρε. Είναι προ δικό του το όφελο, προ το δικό του το μέλλον, για το δικό του το μέλλον που γίνονται όλα αυτά, αλλά και προ το δικό μα το όφελο, διότι έχουμε έτσι την ειρήνη, ε, την ασφάλεια και την σταθερότητα τη παγκόσμια αγορά. Υπ' αυτό το πνεύμα συμφωνώ απολύτω και με όσα είπε η κυρία Γκρέζ με περισσότερες λεπτομέρειες από ό,τι θα αναφέρω εγώ. Ένας φόρος για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές χρειάζεται. Δεν το συμπεριέλαβα αυτό στην συγκεκριμένη έκθεση, γιατί θεώρησα ότι πρόκειται για ένα ευρύτερο μέτρο που δεν αφορά μόνο ε, την αναπτυξιακή πολιτική. ή χρειάζεται να γίνει κάτι τέτοιο για να, να αντιμετωπιστούν οι κλιματικές αλλαγές ή τα αποτελέσματα της τραπεζικής κρίσης. Αυτό που είναι σημαντικό να υποθεί νομίζω είναι ότι Επιτροπή ανέφερε μια σχετική ευελιξία που θα ήταν απαραίτητη όταν μιλάμε για τα κριτήρια της αναπτυξιακής βοήθειας. Όταν σας ακούω να μιλάτε για ευελιξία, και για κριτήρια επιλεξιμότητας πραγματικά φοβάμαι πολύ. Δηλαδή θα δαπανούμε τα κονδύλια μόνο για τα κριτήρια που έχει ορίσει ο ΣΑ και για τίποτε άλλο. Όμως είναι πολύ δύσκολο ήδη να συγκεντρωθούν αυτά τα κονδύλια και κάθε φορά που υπάρχει κρίση κινδυνεύουν τα κονδύλια αυτά τα αποθέματα. Και όποτε υπάρχει ένα πρόβλημα, οι πολίτε μα παρακολουθούν πολύ προσεκτικά πώ δαπανώνται και απαιτούν να δαπανηθούν σωστά. Ε, για σκοπούς δικαιοσύνης λοιπόν και για τις απαιτήσει των πολιτών μας πρέπει να το εξασφαλίσουμε αυτό. Και συμφωνώ, πρέπει να ε, συζητήσουμε, να αγωνιστούμε για τα εργαλεία που διαθέτουμε ώστε να πετύχουμε την κοινωνική δικαιοσύνη, την ισότητα για όλους. Αλλά δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τα ίδια τα κριτήρια. Θα παραμείνω σε αυτά τα σχόλια προ στιγμή. Λυπάμαι που δεν μπορώ να απαντήσω με λεπτομέρειε σε όλα όσα υπόθηκαν. Ήταν νομίζω πολύ χρήσιμη συζήτηση, αλλά επειδή ε, γενικώ ε, συμφωνήσαμε νομίζω, ε, δεν χρειάζεται να μπούμε σε περισσότερε λεπτομέρειε. Πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ. Σα ενημερώνω ότι η ειδική επιτροπή θα ασχοληθεί με τη χρηματοδότηση των εξωτερικών πολιτικών τη Ένωση την 1η Φεβρουαρίου με την παρουσία του Επιτρόπου Πίμπαλξ. Περνάμε τώρα στο σημείο 11 της ημερήσιας διάταξης, μεταναστευτικές ροές που προκύπτουν λόγω της αστάθειας. Πεδίο και ρόλος της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής. Η κυρία Κρετσού έχει ετοιμάσει αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης. Πρόκειται για μια έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και εμείς ζητήσαμε Βάσει του άρθρου 50 να συμμετάσχουμε, να συνεισφέρουμε. Η έκθεση της κυρίας Κατσού είναι πολύ αισιόδοξη διότι μας μιλάει για το φαινόμενο αυτό σαν ένα παράγοντα που μπορεί να βοηθήσει την ανθρώπινη ανάπτυξη. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, θα συνεχίσω στα αγγλικά. Είπατε ότι συνεισφέρουμε σε Επιτροπή στην έκθεση αυτή, Μεταναστευτικέ ροέ που προκύπτουν από την ε, αστάθεια, ρόλο και πεδίο τη Ευρωπαϊκή Εξωτερική πολιτική. Έχουμε εντοπίσει εδώ κάποια ζητήματα και ορίζουμε και κάποιου στόχου μέσω του σχεδίου έκθεση. Απλώ πρέπει να πω ευθύ εξ αρχή ότι ήδη συναντηθήκαμε κάποιε φορέ με τον εισαγητή και του σκεώδει εισηγητέ. Του ευχαριστώ για τη συνεργασία του και τη συμβολή τους, ιδίω την κυρία Κέλλερ, την κυρία, τον κύριο Σφένσον και την κυρία Τσίμερ. Ε, εδώ πρέπει να πω ότι τα κράτη-μέλη σήμερα δεν έχουν ανταποκριθεί με συνέπεια και με σταθερότητα σε ένα φαινόμενο όπως αυτό της μετανάστευσης. Οπότε προσπαθήσαμε με την έκθεση αυτή να συντάξουμε κάποιες συστάσεις ώστε να ενισχύσουμε τις θετικές επιπτώσεις της μετανάστευσης των ε, ανθρώπων Ε, ιδίω σε σχέση με τις μεγάλες ροές από χώρε προέλευσης και την ένταξή τους σε κοινωνίες προορισμού. Συζητήσαμε με την ε, Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για να δούμε κατά πόσο η μετανάστευση μπορεί να προωθήσει την ανάπτυξη στις χώρες μετανάστευσης και τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να μαγιστοποιήσει τα ωφέλη από τις μεταναστευτικές ροές σε περιφερειακό και όλα σε επίπεδο. Βεβαίω, σε κάποια σημεία δεν συμφωνήσαμε με του συναδέλφου τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, όμω επιδιώξαμε συμφωνία ε, στο πρώτο μέρο. Στο δεύτερο μέρο, όπου έχουμε αποκλειστική αρμοδιότητα ω Επιτροπή, έχουμε επικεντρωθεί στον τρόπο κατά τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να βελτιώσει τα ε, μέσα χρηματοδότηση που διαθέτει για την αναπτυξιακή συνεργασία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια ώστε να εξεύρουμε βιώσιμε λύσεις για τους ανθρώπους που ξεφεύγουν από ευάλωτα κράτη. Όπως ξέρετε δεν υπάρχει συμπεφωνημένος κατάλογος ε, με ευάλωτα κράτη. Απλώς ακολουθούμε τις τραπεζικές ταξινομήσεις που εντάσσουν 34 κράτη σε αυτόν τον κατάλογο και 600 εκατομμύρια ανθρώπου που είναι διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο, αλλά κυρίω εντοπίζονται στην Αφρική νοτίω τη Σαχάρα. τη Σαχάρας, μάλλον. Ε, εδώ λοιπόν μιλάμε για χώρε προέλευση και μεταναστευτικά κράτη. Πολλέ φορέ. Έχουμε εκτοπισμένου πληθυσμού, παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κλιματικέ αλλαγέ που οδηγούν στον εκτοπισμό πληθυσμό. Όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία πρέπει να ληφθούν υπόψη για να εξασφαλίσουμε αποτελεσματική προστασία σε αυτού του πολίτε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει δραστικότερα βήματα για να περατώσει τα εργαλεία που διαθέτει στα πλαίσια τη εξωτερική τη δράση και να ενισχύσει τι θετικέ επιπτώσει τη μετανάστευση, προκειμένου να προωθήσει την ανθρώπινη ανάπτυξη και τον εκδημοκρατισμό των ευάλωτων κρατών. Ε, ήδη πέρυσι αγορά της απασχόλησης έχει αποδυναμωθεί σε πολλές χώρες, τις αναπτυσσόμενες, έχουν πέσει τα ποσοστά απασχόλησης στις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες και πολλοί μετανάστες ε, δεν θα επιστρέψουν εύκολα στις πατρίδες τους. Άρα θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες για να μειώσουμε το κόστος των συναλλαγών, να δημιουργήσουμε τέτοιες χρηματοπιστωτικές και οικονομικές συνθήκες, ώστε να υπάρχει διαφάνεια και να εντείνουμε τις σχετικές προσπάθειες. Στο κείμενό μας κάνουμε έκκληση και για στενότερη συνεργασία μεταξύ θεσμικών οργάνων στις αναπτυσσόμενες χώρες και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδώ έχουμε μια σημαντική συνιστόσα την κοινωνία των πολιτών. Επίσης από διεθνούς άποψη, η μετανάστευση μπορεί να γίνει μοχλός για την ενίσχυση του εκδημοκρατισμού και του διαλόγου μεταξύ των ε, κυβερνητικών και μη κυβερνητικών ε, φορέων για την αποστράγγιση την ε, πνευματική ορισμένων χωρών, ιδίω σε ειδικευμένου τομεί. Θα πρέπει να διευκολύνουμε την πρόσβαση ορισμένων ανθρώπων, αλλά με ώστε να αποφύγουμε την κυκλική όπω λέγεται μετανάστευση. Η μετανάστευση είναι πάνω από όλα ανθρώπινα όντα, δεν πρέπει αυτό να το ξεχνάμε. Βεβαίω και έχουν δικαίωμα στα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα, αξιοπρέπεια, ασφάλεια ε, και ειδική προστασία εφόσον απαιτείται. Θα πρέπει λοιπόν ε, μέσω της έκθεσής μας να τονίσουμε ότι τα κράτη-μέλη καλά θα κυρώσουν την Διεθνή Σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των μεταναστών και τα μέλη των οικογενειών τους. Έτσι θα δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο ελάχιστων ανθρωπίνων προτύπων όπως έχουν συμφωνηθεί από την διεθνή κοινότητα ήδη από τη δεκαετία του 1990. Τονίζουμε στην παράγραφο αυτή ότι βασικά ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, διότι πολύ συχνά πολύ εύκολα τα παραβιάζουν ε, οι αρχές του κάτω υποδοχής. για την υπηρεσία εξωτερική δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τι μπορεί να προσφέρει σε όλη αυτή την προσπάθεια και τον ρόλο τη ΔΕΦΚΟ. Εδώ νομίζουμε ότι πρέπει να υπάρξει ε, σταθερό συντονισμό μεταξύ των δύο φορέων και να φροντίσουν να παίξουν έναν αποτελεσματικό ρόλο στην μεταναστευτική μα πολιτική. Και έτσι θα μπορέσουμε να διευκολύνουμε και την επίτευξη των στόχων τη χιλιετία. Θα πρέπει να έχουμε όλες αυτές τις ε, επιδιώξεις υπόψη για την καταπολέμηση της φτώχειας και τις εθνικές αναπτυξιακές στρατηγικές των αναπτυσσόμενων χωρών είναι σημαντικό να δώσουμε ενίσχυση ε, ώστε να αντιμετωπίσουμε μακροπρόθεσμα τα προβλήματα που μας απασχολούν. Σας ευχαριστώ ως τώρα για τις συνεισφορές σας ε, και για τη στήριξή σας. Είμαι πρόθυμη να ακούσω τα σχόλιά σας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Φένσον έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Κρετσού. Είναι πολύ καλή η έκθεση αυτή και θέλω να σας ευχαριστήσω για, την, ε, για το ανοιχτό πνεύμα το οποίο επιδείξατε. Εάν ο κόσμο ήταν ιδανικό, ο καθένα θα πήγαινε όπου ήθελε. Δυστυχώ όμως, καθόλου ιδανικό δεν είναι αυτός ο κόσμος. Κάποιοι πραγματικά είναι υποχρεωμένοι, ξαναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους, τις εστίες τους, τα χωριά τους για λόγους ποικίλου. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Ίσως κάποιες γλωσσικές λεπτομέρειες που τώρα δεν θα τις σχολιάσω, όμως σε κάποια σημεία ήθελα να σταθώ, Πρόεδρε. Παράδειγμα, το σημείο Δέλτα η εισηγήτρια μιλάει για τις θετικές συνέπειες της μετανάστευσης. Πολύ ωραίο αυτό. Όμως, η μετανάστευση πραγματικά δεν πρέπει να θεωρείται ως άχθος για τις χώρες υποδοχής. Έχω όμως μια... έναν ενδιασμό εδώ Δηλαδή η μετανάστευση και ο συσχετισμός της με την ε, ε, μεταρρύθμιση της διακυβέρνηση της χώρας προέλευση. Αυτό είναι σχετικό. Επίση, το σημείο 4. Μιλάμε για τη διασπορά, δηλαδή τους μετανάστες από την ίδια χώρα σε πολλού διαφορετικούς προορισμούς. Εδώ θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η διασπορά έχει δραματίσει και αρνητικό ρόλο. Όπως τη δημιουργία εξτρεμιστικών ε, δικτύων δίκτυα που ενεργούν ή ενεργοποιούνται σε διαφορετικέ χώρε. Το σημείο 10. Παροτρύνουμε όλα τα κάτι μελη τη Ευρωπαϊκή Ένωση να κυρώσουν την ε, Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων όλων των ε, εργαζομένων μεταναστών και των μελών των οικογενειών του. Νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα. Υπάρχει μια δυσκολία. Γιατί Προφανώς και πρέπει να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα όσων ε, μεταναστεύουν για να βρουν δουλειά. Όμως η σύμβαση αυτή είναι πραγματικά αμφιλεγόμενη. Και έχει διατυπωθεί με τρόπο τέτοιο ώστε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην μπορεί να την αποδεχτεί ασυζητητή. Είναι λοιπόν κάπως παράξενο εμείς ως Ευρωκοινοβούλιο να παροτρύνουμε τις κυβερνήσεις μας να κυρώσουν μια σύμβαση που σε κάθε περίπτωση δημιουργεί προβλήματα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Λίβδιν. Νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάποια άλλη διατύπωση. ή να μιλήσουμε για την προστασία των ε, εργαζομένων μεταναστών φροντίζοντας να μην υπάρχουν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Βεβαίως αυτό θα συμπεριληφθεί στις τροπολογίες που θα υποβάλουμε. Επίσης, αναρωτιέμαι κατά πόσον θα πρέπει να μιλήσουμε για τα δικαιώματα των ε, εργαζομένων μεταναστών, ειδικώ εφόσον προέρχονται από πορείες στην Επιτροπή αυτή. Απλώ εμεί θα ζητήσουμε κάποιε μικρέ τροπολογίε. λόγω χάρη τη μετανάστευση λόγω των κλιματικών αλλαγών ή την αναπτυξιακή μα πολιτική και την προσαρμογή τη στη μετανάστευση ή να φροντίσουμε τα κονδύλια που αποδίδονται στην αναπτυξιακή βοήθεια να χρησιμοποιούνται μόνο για αναπτυξιακού σκοπού και όχι για τίποτε άλλο. Αυτό το είχαμε πει και σε προηγούμενη συνεδρίαση. Βεβαίω, η μετανάστευση πολλές φορές ε, οδηγεί σε αυτό το αποτέλεσμα, δηλαδή τα κονδύλια που προσφέρουμε για και βοήθεια να πηγαίνουν και σε άλλα προγράμματα όπως ε, φύλαξη των συνόρων, ε, καταπολέμηση λαθρομετανάστευσης. Αυτό δεν έχει καμία αναπτύξη. Θα πρέπει λοιπόν σαφώς να θέσουμε κάποια όρια και να περιορίσουμε τέτοιες τάσεις. Τα κονδύλια να ε, δαπανώνται για σκοπούς που δεν είναι αναπτυξιακοί. Θα πρέπει αυτό να το εμποδίσουμε. Και συμφωνούμε και για την ε, μνήα της σύμβασης ε, για τα δικαιώματα των εργαζόμενων μεταναστών και των μελών των οικογενειών τους. Σε πολλές περιπτώσεις κάποιοι αναγκάζονται να μεταναστεύσουν γιατί ακριβώς πεθαίνουν από την πείνα, δεν έχουν τρόπο να ζήσουν. Είναι λοιπόν σημαντικό αυτό που αφορά την διεθνή σύμβαση, αυτό που λέγεται για τη διεθνή σύμβαση, γιατί Κάποιες φορές τα βασικά δικαιώματα παραβιάζονται. Δεν είναι λοιπόν μόνο το επιχείρημα των προβλημάτων που έχουν ε, τα κράτη-μέλη μεμονωμένα και για τα παιδιά των μεταναστών κάποιες φορές υπήρξαν προβλήματα. Ε, καθυστερήσαμε και ε, χρονοτριβήσαμε επί χρόνια μέχρι να αποφασίσουμε. αλλά Κάποια στιγμή θα πρέπει να ληφθεί μια απόφαση. Είναι πολύ καλό να αναφέρεται η σύμβαση αυτή στην συγκεκριμένη έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Σνιμπεργιάστρομ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσάς κυρία Κρατού για τη γνωμοδότηση. Στην έκθεσή σας αναφέρεστε γενικά στο θέμα της διαρροής εγκεφάλων, brain drain, αφέμαξη εγκεφάλων. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για την τεράστια σημασία του τομέα της υγείας. Τα τελευταία 30 χρόνια ο αριθμός των ξένων ειδικών επαγγελματιών στον ιατρικό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξανόταν κατά 5% ετησίως από χώρες όπως Αγγόλα, Σιέρα, Λεόνε, Μοζαμβίκη. Περίπου το 60% των εξειδικευμένων εργαζομένων ε, μετανάστευσαν. Αυτή η μετανάστευση έχει τα υπέρ και τα κατά της. Τα πλεονεκτήματα είναι γνωστά, νομίζω. Υπάρχουν τα εμβάσματα που βοηθούν εισοδηματικά, υπάρχει επιμόρφωση των επαγγελματιών αυτών και τα μειονεκτήματα. Ε, πρέπει να τα αναφέρομαι επίσης. Ε γιατί χάνονται τα κονδύλια για την εκπαίδευση ή μετανα... από τη... που έχουν δαπανηθεί στην εκπαίδευση και πολλές φορές ε, δεν μπορούν να ε, εφαρμοστούν συνολικές ε, πρωτοβουλίες για την υγεία, για την αντιμετώπιση του AIDS, της ελονοσίας κλπ. Λείπει ε, λείπουν οι γιατροί που χρειάζονται στις χώρες αυτές. Οι αναπτυσσόμενες χώρες λοιπόν πρέπει να αυξήσουν την ε, ελκτική τους δύναμη προς το επαγγελματικό δυναμικό τους. Αυτό πολλές φορές είναι αδύνατον στην ύπεθρο. Οι επαγγελματίες, οι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τρόπο δικαιότερο, καλύτερο, και θα πρέπει να αμείβονται περισσότερο, το λέμε οι περισσότεροι από εμά, γιατί συνήθως γι' αυτό το λόγο φεύγουν, εγκαταλείπουν τη χώρα τους και πρέπει να ε, ενισχυθεί η εκπαίδευση. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε, να βοηθήσουμε. Πολλές φορές πρέπει να φέρουμε τα παιδιά εδώ για να γίνει η θεραπεία τους. Γιατί να μην ε, εκπαιδεύεται, ε, εκπαιδεύουμε επαγγελματίες της υγείας με προοπτική την επιστροφή τους. Ε, πρέπει λοιπόν να το δούμε και αυτό ως μέρος της προβληματικής της μετανάστευσης και επίσης να έχουμε και ένα παγκόσμιο κώδικα δεοντολογία στον τομέα αυτό, όπως ε, προβλέπεται και από τον ΠΟΕ. Να δούμε δηλαδή συνολικότερα το θέμα. Ο κύριος Μαρτίνες. Ευχαριστώ κι εγώ. Αυτά που μας παρουσίασε η κυρία Κρέτου είναι σωστά. Τη συγχαίρω. Μου λείπει όμως ένα στοιχείο διεξόδου. Μια προοπτική ιστορική σημασίας που λείπει πρέπει να πούμε ότι όλες οι χώρες μας, χωρίς εξαίρεση, είναι χώρες που έχουν παράδοση μετανάστευσης από τη χώρα προς τα έξω. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι η Σουηδία, που ήταν μοντέλο για τους ανθρώπους της γενιάς μου όσον αφορά την πρόοδο και τα λοιπά, ότι κάποια στιγμή έγινε η χώρα της Ευρώπης που είχε περισσότερη θυματίωση, περισσότερη ανεργία και μένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό ε, ανθρώπων που έφευγαν με πλοία και πηγαίνανε στην Αμερική ή πηγαίνανε στην Αργεντινή. Πόσοι Σουηδοί δεν έχουν πάει στην Αργεντινή. Αυτή είναι πραγματικότητα πιο σύγχρονη για την Ισπανία. Η Ισπανία δεν είχε μόνο 3-4 εκατομμύρια ανθρώπων που έφυγαν από την Ισπανία και πήγανε στη Λατινική Αμερική, αλλά είχε και πάρα πολλούς που πήγανε σε ευρωπαϊκές χώρες, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λουξεμβούργο. Εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια Ρουμάνοι είναι σε ευρωπαϊκές χώρες. Ένα εκατομμύριο έχουμε στην Ισπανία Ρουμάνους μετανάστες, οι οποίοι μετανάστευσαν από τη χώρα τους προς την Ισπανία στην Ρουμανία μπορεί να το ξέρουν. Γιατί όλοι έχουν συγγενείς στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Ισπανία. Όμως κανένας νέος Ισπανός ή παιδί Ισπανός δεν ξέρει ότι εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτε του αναγκάστηκαν κάποια στιγμή και φύγανε και πήγανε στη Γερμανία, στην Αγγλία ή αλλού. Και πότε, πριν από 30 χρόνια, ε. δεν μιλάω για πολύ πιο παλιά. Οι νέοι δεν μπορούν να το διανοηθούν ότι οι άνθρωποι έπρεπε να φύγουν από τη χώρα τους για να βρούνε το ψωμί τους, να μπορέσουν να φάνε. Αυτή λοιπόν είναι μια ιστορική πραγματικότητα. Οι χώρες μας κατά παράδοση ήταν χώρες που επηρέαστηκαν πάρα πολύ από τη μετανάστευση αλλά με δημοκρατικούς μηχανισμούς, με μηχανισμούς σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κοινωνικής δικαιοσύνης, κατάφεραν να ανατρέψουν την τάση. Και οι χώρες μας υποδέχονται πια μετανάστες. Και δεν είμαστε εμείς που μεταναστεύουμε προς άλλες χώρες. Αυτό μου λείπει από την έκθεση. Θα ήθελα κάπου να αναφέρετε. Θα μου άρεσε να το δω στην έκθεσή σας, κυρία Κρετού. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κορτές Γάστρα τώρα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ την εισηγήτρια για τη δουλειά της, για την γνωμοδότησή της και συμφωνώ απόλυτα με τον Μιγελάχελ αυτό που είπε. Ότι θα ήταν πολύ καλό κάπου να γίνεται μια ιστορική αναδρομή. Να δούμε τι είχε γίνει πριν εκατομμύρια φύγανε από την Ισπανία προς την Ευρώπη κάποια στιγμή. Την Ιρλανδία επίσης. Ή από την Ευρώπη προς άλλες χώρες του κόσμου. Αυτό πρέπει να φαίνεται, να είναι οπτό. Τώρα θα είμαι σύντομος, κύριε Πρόεδρε, για την έκθεση αυτή καθ' αυτή. Σημερίζομαι τρεις από τις ιδέες που αναφέρει η συγγήτρια και θέλω να σχολιάσω σε αυτές. Πρώτον, ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε τις αιτίε που οδηγούν στη μετανάστευση. Δεύτερον, να μειωθεί το κόστος που έχουμε σήμερα εξαιτία της ε, μετανάστευσης αυτής. Να καταπολεμηθούν δηλαδή αίτια όπως είναι η φτώχεια. Και να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο της διαφυγής εγκεφάλων. Υπάρχουν νέες χώρες που αναδύονται και πια οι επιστήμονες δεν φεύγουν μόνο προς τις Ηνωμένε Πολιτείες, πάνε και αλλού. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος και είναι κρίμα. Εμείς θέλουμε ανάπτυξη, έρευνα, καινοτομία, το να αφήνουμε τους ανθρώπους να φεύγουν και να πηγαίνουν ε, αλλού είναι κρίμα. Και επιμένω στην σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη μετανάστευση και την ανάπτυξη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριλάβει τη μετανάστευση σαν ένα εγκάρσιο στοιχείο σε όλες τις, τις στρατηγικές για την ανάπτυξη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκέρενς τώρα. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστούμε ιδιαίτερα την κυρία Κρατού που ξεκίνησε τη συζήτηση. Έχω απλώς δύο απορίες. Πρώτον, στο σημείο 16 χαιρετίζεται τη δημιουργία του παρατηρητηρίου για τη μετανάστευση. Αναρωτιέμαι, δεν υπάρχουν ήδη αρκετά παρατηρητήρια και της Αφρικανικής Ένωσης. Χρειάζεται και ένα παρατηρητήριο ΑΚΕ. Δεν ξέρω, ερώτηση είναι. Αλλά Καλό θα ήταν να κάνουμε πρώτα και μια συνολική εξετάση των, του πόσα παρατηρητήρια ήδη υπάρχουν. Και ένα ακόμη ερώτημα προς τον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Όταν βρίσκεστε σε διαπραγματεύσεις για θέματα μετανάστευσης με τρίτες χώρες, διαπραγματεύεστε με την κάθε χώρα ξεχωριστά ή με τις χώρες ομαδικά όπως ε, οι χώροι ελεύθερων συναλλαγών που έχουν δημιουργηθεί. Διότι αν το σκεφτεί αυτό κανεί σε σχέση με τι χώρε τη Δυτική Αφρική λόγου χάρη, είναι διαφορετικό από το να διαπραγματεύεται κανεί ξεχωριστά με την κάθε χώρα όπω τη Σενεγάλη, το Μαλί και το καθεξή. Εμεί έχουμε δημιουργήσει ένα τέτοιο χώρο ελεύθερων συναλλαγών συζητούμε συμφωνίες που συλλογικά, πράγμα που μεταμορφώνει ουσιαστικά το πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του χώρου του Σέγγεν. Θα ήθελα λοιπόν εδώ κάποια ε, διευκρίνηση και μια τρίτη παρατήρηση, να στηρίξω πλήρως όσα είπατε κι εσείς, για την διαφυγή των εγκεφάλων των επιστημόνων από τις τρίτες χώρες προτείνατε να δώσουμε τέτοιες δυνατότητες στους γιατρούς λόγου χάρη που να μπορούν να εκπαιδευτούν στις χώρες μας και να επιστρέφουν μετά στη δική τους. Όμως, από τη μια θα πληρώνουμε υποτροφίες των φοιτητών από αναπτυσσόμενε χώρες. Από την άλλη, πρέπει να του ζητήσουμε τουλάχιστον να εκτίσουν μια να, θητεία στη χώρα προέλευση του Για ένα ελάχιστο διάστημα. Και το λιγότερο μπορούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε θεωρήσεις πολλαπλών εισόδων στους ε, Αφρικανούς πολίτες, οι οποίοι επιθυμούν να έρθουν στην Ευρώπη για να συμπληρώσουν την εκπαίδευσή τους. Υπάρχουν προγράμματα δημοποίησης και υπάρχουν εμπειρογνώμονες που θα ενδιαφέρονταν. Καλό θα ήταν να υπάρχει λοιπόν ένα τέτοιο σύστημα που να επιτρέπει το πηγενέλα μεταξύ χωρών προέλευσης και Ευρωπαϊκής Ένωση. Ευχαριστούμε. Υπάρχει κάποιος στην αίθουσα από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Όχι. Ξαναδίνω το, το, λόγο στην κυρία Κρατσού για να ολοκληρώσει. Thank you very much Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Από ευθύς εξ αρχής να πω ότι γιατί στη διαδικασία κατάρτισης του σχεδίου της νομοδότησης το πιο δύσκολο ήταν να καλύψω και να αναφέρω όλα τα θέματα που επηρεάζονται γιατί έχουμε περιορισμένο χώρο και η μετανάστευση ε, πρέπει να καλύψει πολλά θέματα. Επίσης, είναι μόνο γνωμοδότηση η δική μας, η άφετη αρμόδια, ε, σκοπός και ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, πολιτική μεταναστευτικών ε, ρευμάτων που οφείλονται στην αστάθεια είναι ο τίτλος. Ευχαριστώ όμως για όλα τα σχόλια, όλες τις παρεμβάσεις σας. Τώρα, για τον κύριο Σβένσον. Στη δεύτερη παράγραφο αναφερθήκατε εσείς ε, η μετανάστευση και η ανάπτυξη είναι διασυνδεδεμένα φαινόμενα. Λέμε εκεί και τονίζουμε τα θετικά της μετανάστευσης που μπορούν να συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη, την οικονομική μεγέθυνση, την κοινωνική ενίσχυση, την τεχνολογική πρόοδο και καμιά φορά και σε μεταρρυθμίσεις. Είσαστε στις συζητήσεις που κάναμε με προσώπους της ΑΦΕΤ. Στο κείμενο έλεγε ότι καμιά φορά η μετανάστευση είναι και πηγή τρομοκρατίας και εμείς ε, ως ΔΕΒΕ δεν θέλαμε αυτή τη γενίκευση με βάση κάποια μεμονωμένα περιστατικά ήταν λοιπόν σκληρές οι διαπραγματεύσεις για το κείμενο με τους εκπροσώπους της ΑΦΕΤ για να δείξουμε τα θετικά της μετανάστευσης και όχι μόνο τις αρνητικές επιπτώσεις. Βέβαια, η διασπορά θεωρώ ότι είναι σημαντική συνιστόσα οποιασδήποτε κοινωνία των πολιτών. Πολλές χώρες στην Ευρώπη, δεν ξέρω για τη Σουηδία, αλλά σε πολλές χώρες της Ευρώπης η διασπορά παίζει σημαντικό ρόλο. Και ο στόχος μας ήταν όχι να απομονώσουμε τις ομάδες της διασποράς, αλλά να τις εντάξουμε στην κοινωνία. Για τους εργαζομένους, βέβαια αυτό είναι ένα θέμα πολύ αμφιλεγόμενο, η προστασία των εργαζομένων και το δικαίωμα εργασίας ιδιαίτερα τώρα με την κρίση όπου πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν γίνει πιο εγωιστικές στην πολιτική τους, αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει να τονίσω με το δικαίωμα αυτών των ανθρώπων να έχουν μια θέση απασχόλησης και το δικαίωμά τους να εντάξουν και την οικογένειά τους στη νέα χώρα. Επίσης χαιρετίζω ιδιαίτερα την παρέμβαση της κυρίας Κέλλερ η οποία υπογράμμισε την ιδέα της μετανάστευσης ως ανθρώπινο δικαίωμα. Πολύ ε, εκτιμώ την συμβολή της σε αυτό το θέμα της προαγωγής της κινητικότητας, ε, αυτή την αναγκαστική επιλογή και την αναφορά της ανθρώπινα δικαιώματα γιατί ήταν εισηγήτρια ε, από την Επιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κυρία Σνάιμπερ, συγγνώμη αν δεν το λέω σωστά το όνομά σας, αυτός, αυτή η αφέμαξη εγκεφάλων είναι πολύ σημαντικό θέμα, ιδιαίτερα στην ιατρική. Ιδιαίτερα αφορά αυτό την Αφρική. Πολλοί Αφρικανοί φεύγουν Βεβαίως τα εμβάσματα είναι πολύ σημαντικά για τη χώρα από τους ανθρώπους αυτούς, από την άλλη μένουν χωρίς ειδικού. Γι' αυτό μιλάμε και για την κυκλική μετανάστευση όπου φεύγουν, έρχονται, ξαναφεύγουν, είναι επιλογή αυτών των ανθρώπων και δεν μπορούμε να είμαστε κατά όπως είπε και ο Μιγγέλ, όπως είπε και ο κύριος Μαρτίνες στη δική του παρέμβαση, αυτό το πρόβλημα υπάρχει και στην Ευρώπη. Η Ρουμανία έχασε πολλούς ειδικού επαγγελματίες. Δεν φεύγουν μόνο οι τσιγκάνοι, αλλά και πολλοί καθηγητές, γιατροί, οπότε αυτό αποτελεί απώλεια για τη χώρα. Πάντως, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αν οι άνθρωποι αυτοί επιλέξουν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους και να αναζητήσουν καλύτερη ζωή αλλού, πρέπει να ενθαρρύνουμε τις επιλογές τους και να τους προσφέρουμε κάποιες ευκαιρίες στη χώρα που επιλέγουν να εγκατασταθούν. Παράλληλα, βέβαια, θα πρέπει, ιδιαίτερα στις πολύ φτωχές χώρες, όπως είναι οι αφρικανικές, πρέπει να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να επιστρέφει. Αλλά οι κυβερνήσεις που έχουν τέτοιο χαμηλό επίπεδο και οικονομική ανάπτυξη δεν μπορούν να τους προσφέρουν τους ίδιους μισθούς όπως έχουν στις Βρυξέλλες ή στη Γαλλία ή οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη. Οπότε εκείνοι επιλέγουν ποια θα είναι η ζωή τους. Αυτές είναι οι επιλογές ζωής. Επίσης υπάρχει το θέμα των περιορισμών στην αγορά. από τις δυνάμεις της αγοράς. Και αυτό το συζητήσαμε με τους συναδέλφους από την Επιτροπή Απασχόλησης, δηλαδή την μπλε κάρτα ε, για την προσέλκυση ειδικών, αλλά και την ε, δυνατότητα να μπλοκάρουμε μερικούς. Ο κ. Γκέρενς μίλησε για το ε, μεταναστευτικό μηχανισμό για τις χώρες ΑΚΕ. Αυτό άρχισε να λειτουργεί από πέρσι τον Οκτώβριο. Πέρσι δηλαδή δημιουργήθηκε και βέβαια το χαιρετίζουμε γιατί ο βασικός στόχος αυτού του μεταναστευτικού μέσου για τις χώρες ΑΚΕ είναι να βοηθήσει στη διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων στα σύνορα των χωρών και Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πολλά ακόμα μπορεί κανείς να πει για τη μετανάστευση και τις επιπτώσεις του φαινομένου αυτού, αλλά υπενθυμίζω επίσης ότι έχουμε μία προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Όλοι παρακαλείστε να συμβάλλετε στην έκθεση αυτή. 1η Φεβρουαρίου είναι η προθεσμία και η ψηφοφορία στην Επιτροπή θα είναι 3 Μαρτίου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 12 της ημερήσιας διάταξης, μελλοντική ευρωπαϊκή πολιτική για τις διεθνείς επενδύσεις. Είναι έκθεση που ετοιμάζει η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και επειδή Υπάρχουν βεβαίω, προφανείς συνέπειε για την ανάπτυξη. Η δική μα Επιτροπή ετοιμάζει γνωμοδότηση. Ο κύριος Μπιλ Νιούτον Ντάν είναι υπεύθυνο για αυτήν την έκθεση. Του δίνω το λόγο για να μα παρουσιάσει αυτά που ετοιμάζει. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αυτή είναι μια γνωμοδότηση της ΣΥΝΤΑ που έχουν καταρτήσει και έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας ως αποτέλεσμα της ε, θέσης σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνα, στη Λισαβόνας, η οποία δίνει αποκλειστική αρμοδιότητα στην Επιτροπή στην Διεθνή Επενδυτική Πολιτική της Ένωσης και την δυνατότητα να καταργεί τους περιορισμούς στην Εθνική Επενδυτική Πολιτική. Η γνωμοδότηση αυτή που συνέταξα για σας δίνει ε, τη γνώμη της Επιτροπής μας στην ΙΝΤΑ σχετικά με την αναπτυξιακή πλευρά της διεθνούς επενδυτικής πολιτικής, γιατί η έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας της ΙΝΤΑ και η ανακοίνωση της Κομισιόν επί του θέματος είναι πολύ πιο γενικές και αφορούν τις αναπτυγμένες χώρες και λιγότερο τις ε, αναπτυσσόμενες. Α, με βοηθάει ο κύριος ε, Μπέρμαν. Να συνεχίσει να με βοηθάς. Ε, λοιπόν, ε, έχω... η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι αύριο το βράδυ. Υπάρχει χρόνος δηλαδή να καλάξετε τις προτάσεις με αυτό που με απογοητεύει είναι ότι η ανακοίνωση της Κομισιόν πολύ λίγο χρόνο θα πανά στις αναπτυσσόμενες χώρες ε, ως δυνητικούς επενδυτικούς εταίρους και επικεντρώνται κυρίως στις μεγάλες αγορές του κόσμου. Πρέπει να θυμίσουμε στην Κομισιόν, η Ίντα να το θυμίσει, ότι η συνθήκη ε, υποχρεώνει την ε, Ένωση να κάνει συνεκτική πολιτική για την ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη των στόχων στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς επηρεάζουν τις αναπτυσσόμενες χώρες. Διάφορα θέματα θέλουμε να συμπεριλάβουμε, όπως ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για το περιβάλλον, για συνθήκες εργασίας, για τη διαφάνεια και τις παράνομες κεφαλαιακές ροές. Θέλουμε λοιπόν να ζητήσουμε από την Ίντα να ε, συμπεριλάβει θέματα δημιουργίας ικανοτήτων, διακυβέρνησης, για τη δικαστική εξουσία, το κοινοβούλιο, τις υποδομές, την ενίσχυση του φορολογικού συστήματος, την πρόθεση της πρόσβασης στα κεφάλαια και στις μικροπιστώσεις, ε, σύμφωνα με την πρόσφατη πράσινη βίβλο της ε, Κομισιόν για την Αναπτυξιακή Πολιτική και θέλουμε ήταν να αναγνωρίσει τη σημασία των ίσων όρων του παιχνιδιού. Να θυμάται όμως ότι υπάρχουν τεράστιες ανισορροπίες μεταξύ ορισμένων εύθραυστων αναπτυσσομένων οικονομιών. Και έτσι η αμοιβαιότητα θα πρέπει ίσως να διαφοροποιείται σε ορισμένες περιπτώσεις. Οπότε, αν και πιστεύω ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες θα ωφεληθούν πολύ, αν είναι ενιαίος ο συνομιλητής η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις επενδύσεις και να μην είναι μόνο επιμέρους συμφωνίες με τις χώρες των 27, θα ήθελα να ζητήσω από την Ίντα να συμπεριλάβει τα θέματα αυτά στην ε, εκθεσή της. Προσπάθησα να είμαι σύντομος, κυρία Πρόεδρε, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Με ενδιαφέρει η γνώμη των συναδέλφων. Μπορούμε να προτείνουμε τροπολογίε να καταθέσουμε μέχρι το βράδυ και η πρόταση είναι να γίνει ψηφοφορία στην Επιτροπή μας στις 7 Φεβρουαρίου. Η κυρία Κέλλερ ευχαριστώ. Η Τζούντιθ Αργεντίνη ήταν η σκιώδη την αντικαθιστώ και θα πω τις παρατηρήσεις της και τις δικές μου. Συγκεκριμένα, δεν είμαστε βέβαιοι, απόλυτα βέβαιοι, αν η εξίσωση επενδύσεων ανάπτυξης και μεγέθυνσης είναι πάντα τόσο σαφής και αν είναι σωστό να τα εξισώνουμε αυτά τα τρία γιατί η ανάπτυξη είναι στόχος. Ε, διερεύνηση θεμάτων, ελευθεριών, ανθρωπίνων δικαιωμάτων κλπ. Η μεγέθυνση δεν είναι καθ' αυτό στόχος. Επίσης, η επένδυση που αναγκαστικά οδηγεί στην ανάπτυξη, ε, δεν είναι πάντα η διασύνδεση αυτή τόσο σαφής, γιατί η ανάπτυξη ποιον θα, δηλαδή, ποιον θα ωφελήσει, τον τόπιο πληθυσμό, την εταιρεία που επενδύει, ποιον θα ωφελήσει και τι είδου ανάπτυξη θα δημιουργηθεί. Μπορεί η επένδυση να οδηγήσει σε ανάπτυξη, αλλά αυτό δεν είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη προϋπόθεση. Επίσης, το 1998, πέρασαν πολλά χρόνια από τότε, αλλά θα πρέπει να το δούμε, έγινε μια ανάλυση, μια έκθεση τότε και είδαμε ότι υπάρχει πολύ μικρή σχέση μεταξύ ε, επενδυτικών συμφωνιών και αλλαγές στις ροές του αναπτυξιακού μέσου για τη συνεργασία. Επίσης το όλο θέμα της αντιμετώπισης των ξένων εταιριών και η αντιμετώπιση τους ως εθνικών. Πάλι εδώ δεν είναι ίση όρη του παιχνιδιού γιατί οι ξένοι επενδυτές έχουν κάποια προνόμια που δεν τα έχουν οι εθνικοί επενδυτές. Αν δηλαδή έχουν και εθνικά δικαιώματα οι ξένοι επενδυτές και τα προνόμια των ξένων, αυτομάτως ε, αλλάζουν, διαστρεβλώνονται οι όροι του παιχνιδιού. Εάν θέλουμε να έχουμε επενδύσεις επιτόπου να λειτουργούν, πρέπει να τα δούμε όλα αυτά και να μην το παρακάνουμε με τα προνόμια που προσφέρουμε στους ξένους επενδυτές και μετά να μιλάμε για ίσους κανόνες του παιχνιδιού. Ε, ο ΣΑ λέει ότι θέλουν ίσες ευκαιρίες, δηλαδή όχι να δίνονται προνόμια στους ξένους επενδυτές. Επίσης κάτι που με εντυπωσιάζει πάντα στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών είναι το θέμα των απαλωτριώσεων ή και των έμεσων απαλωτριώσεων. Αυτό δεν το αναφέρετε από ό,τι βλέπω στη γνωμοδότησή σας και θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας για αυτό το θέμα ότι χώρες μπορεί να χρειαστεί να καταβάλουν αποζημιώσει για κάτι που λέγεται έμεσε απαλωτριώσει, που δεν είναι καθ' αυτό απαλωτρίωση, αλλά αν η χώρα λάσει με τον περιβαλλοντικό της νόμο και ο επενδυτή κληθεί να πληρώσει για νέα πρότυπα, αυτή είναι μια έμεση απαλωτρίωση ή τις απεργίες κλπ. Μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που εμπίπτουν στον ορισμό του ε, τη έμεση απαλωτρίωση. Αυτό είναι επικίνδυνο, ιδιαίτερα βλέποντα τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Αλλά υπάρχουν και άλλοι τομεί προβληματικοί εδώ. Καλό θα ήταν λοιπόν να ασχοληθείτε με το θέμα. Τι σκέψεις κάνετε ή μήπως καταλήγετε σε διαφορετικά συμπεράσματα από τη μελέτη σας, ε, από τα δικά μου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκούρενς. Μια ερώτηση. Έχει τόσο προ τον εισηγητή, τον οποίο συγχαίρω γιατί τόσο ενδιαφέρουσα παρουσίασή του, αλλά η ερώτησή μου έχει να κάνει με τις εξωτερικές πτυχές της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο εισηγητής πολύ σωστά είπε ότι όσον αφορά την ε, επενδυτική πολιτική μας, ότι είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συμπεραίνω ότι η υπηρεσία εξωτερικής δράσης δεν είναι αρμόδια για το θέμα. Παρ' όλα αυτά, για λόγους συνοχής της εξωτερικής μας πολιτικής, θα ήθελα να γνωρίζω υπάρχει ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα ε, στους υπεύθυνους της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης και των υπηρεσιών αντίστοιχα αρμόδιων ε, για αυτά τα θέματα από την Επιτροπή. Και από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ποιο κάνει τι διαπραγματεύσει για συμφωνίε που προωθούν τι διευκολύνσει στον τομέα των επενδύσεων. Ποιο είναι υπεύθυνο για αυτή την πολιτική. Στην πράξη δηλαδή, πώς γίνεται. Θα ήθελα επίσης οι εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Εξωτερικών Δράσεων να με ενημερώσουν για τις διαδικασίες που ακολουθούν και με ποιο τρόπο η υπηρεσία αυτή εμπλέκεται στις διαδικασίες. Ο κύριος Κορτές Γάστρη, το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγχαρητήρια στον εισηγητή, τον κύριο Νιούτον, για το έργο του. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα των επενδύσεων και είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι χρειάζεται μια ευρωπαϊκή πολιτική για τις επενδύσεις που να είναι συνεκτική και να συνάδει με τις αρχές μας όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Θέλω να ξέρω πιο συγκεκριμένα όμως πώς λαμβάνεται υπόψη η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Και θέλω και να υπογραμμίσω το ρόλο που μπορούν να παίξουν οι ευρωπαϊκές επενδύσεις στην μεταφορά τεχνολογίας κυρίως όταν πρόκειται για τις πράσινες τεχνολογίες. Πρέπει επίσης να υπάρχει και μία κοινωνική ευθύνη που να συνοδεύει τις επενδύσεις αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ θερμά, Πρόεδρε. Κατά πρώτον ευχαριστώ τον συγητή, τον κύριο Νιούτον Ντάν, για την έκθεσή του και να πω ότι θα συμφωνήσω με τις ανησυχίες της Επιτροπής μας για όλη αυτή την θεματική που σχετίζεται με τη μελλοντική επενδυτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να υπογραμμίσω ότι θα συμφωνήσω με τις ανησυχίες που εκφράζει η έκθεση, διότι για την ώρα δεν έχει ληφθεί υπόψη η κατάσταση των αναπτυσσόμενων χωρών στα πλαίσια των ολοδιαπραγματεύσεων. Να θυμίσω με τη σειρά μου ότι η συνεκτικότητα των αναπτυξιακών πολιτισμών, πολιτικών συγγνώμη, είναι κάτι που προβλέπει η ίδια συνθήκη. Χρειάζεται λοιπόν μεγαλύτερη προώθηση των επενδύσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες, κάτι απαραίτητο και ωφέλιμο και για τις ίδιες αυτές τι αναπτυσσόμενε χώρε. Πρέπει όλα αυτά γίνουν με ένα βαθμό ευελιξία ώστε να προσελκύσουμε του πλέον κατάλληλου για την κάθε χώρα επενδυτέ και οι οποίοι είναι σε θέση να προσφέρουν βιώσιμη ανάπτυξη χάρη στι βοήθειέ του. Επίση, είναι καθοριστική σημασία να εμβαθύνουμε την ε, συνεργασία στην αναπτυξιακή βοήθεια για να βελτιώσουμε τη θεσμική, το θεσμικό συντονισμό και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην αγορά τέλος δεν αρκεί να προωθήσουμε τις επενδύσεις στις αναπτυσσόμενε χώρες μόνον, αλλά θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι και οι τοπικές επιχειρήσεις ε, την χάνουν στήριξη για να βεβαιωθούμε ότι πραγματικά ωφελούνται από τι ξένε επενδύσεις. Νομίζω ότι η ομάδα του ΕΛΚ θα μπορέσει να υποβάλει τροπολογίες ε, εμβαθύνοντας και προωθώντας τις κατευθύνσεις που σας ε, περιέγραψα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε η Επιτροπή τώρα με τον κύριο Μαραγκόνη. Με συγχωρείτε μια μικρή αλλαγή. Εδώ έχουμε τον κύριο Ρουπινάτσι από την Γενική Διεύθυνση Εμπορίου που θα παρέμβει. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους βουλευτές για τις χρήσιμες ενισφορές τους. Δύο-τρεις παρατηρήσεις μόνον. Κατά πρώτον, η ανακοίνωση αυτή αφορά κυρίως την έναρξη πολιτικής συζήτησης για το ποιες είναι οι νέες αρμοδιότητες. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε την ανακοίνωση αυτή πιστή σε ορισμένες μέρημνες, αλλά και αρκετά ανοιχτή, ώστε να συγκεντρώσουμε και να συλλέξουμε τις απόψεις των διαφορών ε, ενδιαφερομένων. Σε σχέση με την επιλογή εταίρων τρίτων χωρών με τους οποίους να διαπραγματευτούμε επενδυτικές συμφωνίες. Θεωρούμε ότι η είναι αρκετά ευρεία στην προσέγγιση της και προβλέπει και ένα ευρύ σύνολο κριτηρίων. Αληθεύει ότι βραχυπρόθεσμα προτείναμε να ξεκινήσουμε με κάποιες χώρες με τις οποίες ήδη υπάρχουν ε, διπλωματεύσεις εξέλιξη. Ωστόσο, τα κριτήρια που προτείνουμε για τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δράσεις μας νομίζουμε είναι αρκετά ανοιχτά, ώστε να επιτρέψουν και σε άλλες αναπτυσσόμενες χώρες να συμμετάσχουν. Ε, πραγματικά μπορείτε να είστε ήσυχοι ότι βλέπουμε την ανάγκη αυτή των αναπτυσσόμενων χωρών να συμμετάσχουν σε αυτές τις ε, ε, Συζητήσει όταν αναζητούμε μελλοντικού εταίρου. Επίση, για τα σχόλια που αφορούν την ε, συνοχή την πολιτική. Νομίζουμε ότι και αυτό είναι πολύ σημαντικό και η κοινή ε, επενδυτική πολιτική ω μέρο τη κοινή εμπορική πολιτική θα πρέπει να καθοδηγείται από τι αρχέ και του στόχου τη ευρωπαϊκή εξωτερική δράση, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων όπω η προώθηση του κράτου δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη βιώσιμη ανάπτυξη. Βεβαίω, είναι σαφέ ότι οι μελλοντικέ επενδυτικέ συμφωνίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι συνεπεί και με τι άλλε πολιτικέ που έχουμε σχεδιάσει. Αναγνωρίζουμε ότι θα υπάρξει ανάγκη να έχουμε τη σωστή ισορροπία από τη μια με το, το δημόσιο συμφέρον και τις κρατικές πολιτικές αλλά και την προστασία των ξερών επενδυτών στο εξωτερικό από την άλλη. Νομίζουμε ότι αυτά είναι σημαντικά σημεία. Σε ό,τι αφορά την όλη συζήτηση για τις προδιαγραφές προστασίας, είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Θα φροντίσουμε να εμβαθύνουμε. Και τέλος, για να απαντήσω στον κύριο Γκέρενς, ο Επίτροπος Εμπορίου έχει αναλάβει την εξέταση αυτών των συμφωνιών ε, με βάση τις κατεντήριες γραμμές που ενέκρινε το Συμβούλιο Προφανώς εδώ θα καλύπτονται και οι μηχανισμοί συντονισμού και με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα, όχι, ο κύριος Νιούτον Ντάν έχει το λόγο για να ολοκληρώσει. Γρήγορα, πολύ σύντομα, επειδή πέρασε η ώρα, πάρα πολλά και πολύ επικοδομητικά σχόλια. Ευχαριστώ όλους. Δεδομένε τη λήξη τη προθεσμία αύριο τέτοια ώρα, κάποιοι συνάδελφοι, όχι, έφυγε ο συνάδελφο από το ΕΛΚ, αλλά υποσχέθηκε τροπολογίε. Τέλο πάντων, θα έλεγα σε όσου δεν έχουν χρόνο να προσπαθήσουν να υποβάλουν προφορικέ τροπολογίε για να φτάσουν όλα αυτά στι πληροφορίε. Βρίσκω τα σχόλια πολύ θετικέ συνεισφορέ. Αν λοιπόν γίνουν προφορικέ τροπολογίε υπό το πνεύμα τη συζήτηση που μόλι κάναμε, ευχαρίστω να τη στηρίξω. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Θυμίζω, όπω είπε ο κ. Νιωτοντάν, ε, υποβολή τροπολογιών ω αύριο στι 5. Και θα ψηφίσουμε στην ερχόμενη συνεδρίασή μα τον Φεβρουάριο. Τώρα, σημείο 14 τη ημερήσια διάταξη, Θα θυμάστε ότι το 13 το αναβάλαμε για αύριο, επειδή έλειπε ο κ. Δέβα. Οπότε, Έχουμε τώρα τη γνωμοδότησή μας για το πρωτόκολλο που ορίζει αλληλευτικές δυνατότητες και, ε, και χρηματικά, οικονομικά μάλλον για τον τομέα της αλίας και τη σχετική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και νησών Κομορών. Κάποιοι από εσά θα πρέπει να θυμούνται τη συζήτηση που είχαμε κάνει σχετικά με τις αλληλευτικές συμφωνίες με τις Κομόρες και με τη Γουινέα Κόνακρη και οι εμπειρογνώμονες που είχαν προσκληθεί μας παρουσίασαν πολλά σχετικά στοιχεία. Είχα εκφράσει εγώ μια πολύ σαφή άποψη για το γεγονός ότι οι συμφωνίες αυτές δεν μπορούν να θεωρούνται ως συμφωνίες που έχουν σχέση με την ανάπτυξη. Όμως δεν τα αποφασίζουμε εμείς αυτό έτσι κι αλλιώς. Δεν αποφασίζουμε εμείς για τις ελληνικές συμφωνίες, αλλά η Επιτροπή Αλίας. Θα πρέπει λοιπόν να ετοιμάσουμε γνωμοδότηση η οποία ενδεχομένως να καλυφθεί από την καθήλυνα αρμόδια επιτροπή. Σας θυμίζω ότι η συμφωνία αυτή με τις Κομόρες ε, αφορά τη δυνατότητα 70 σκαφών να αλλιεύουν 4.850 τόνους με αντάλλαγμα 1.845.000 845.000 ε, περίπου ευρώ. Αυτό ισοδυναμεί με 65 ευρώ τον τόνο. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι μου φαίνεται γελίο το ποσό αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλει 300.000 ευρώ για την στήριξη της τομεακής αλληλευτικής πολιτικής των Κομορών. Η απονομή των κονδυλίων αυτών είναι ένα ευαίσθητο σημείο και θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι τα χρήματα αυτά πηγαίνουν πραγματικά στις κοινότητες των ψαράδων στις Κομόρες και δεν καταλήγουν στους κατα... στις τσέπες των διεφθαρμένων πολιτικών εθνών πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε από την Επιτροπή Αλίας να συμπεριλάβει στην έκθεσή της απαιτήσει, συγκεκριμένε απαιτήσει και όρου ό,τι αφορά την διαφάνεια των διαδικασιών που επιτρέπουν να καταγράψει κανείς το σύνολο των τελικών αλλιευμάτων, διότι έχουμε δει από άλλες εμπειρογνωμοσύνες αλλού ότι υπάρχουν σοβαρές απώλειες συνήθως. Επίσης να βεβαιωθούν και την εντιμότητα και την χρηστή ε, χρησιμοποίηση των μηχανισμών λόγω του φαινομένου της διαφθοράς. Αυτό είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο, διότι ξέρουμε ότι δεν έχουμε πετύχει ως τώρα πολλές τέτοιους τομείς και πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι τοπικές κυβερνήσεις που σκοπό έχουν να βελτιώσουν τη διαβίωση των ψαράδων και των τοπικών κοινοτήτων τους, όλα αυτά θα ενισχυθούν. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν με 300.000 ευρώ. Ενώ αν δεν πηγαίναμε να λιεύσουμε εκεί, δεν θα χρειαζόταν να βελτιώσουμε τίποτα. Δεν θα πειράζαμε καθόλου τους τοπικούς ψαράδες. Θα πρέπει λοιπόν να πετύχουμε σε τακτική βάση να μας αποστέλλονται εκθέσεις για την υλοποίηση μιας τέτοιας συμφωνίας. Αυτά. Να σας δώσω το λόγο. Η κυρία Κέλλερ έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με όσα είπατε και ήθελα να κάνω μια γενικότερη παρατήρηση για τις αλληλευτικές συμφωνίες. Αφότου το Ευρωκοινοβούλιο έχει αρμοδιότητα συναμόφασης, μάλλον την ε, διαδικασία της σύμφωνης γνώμης, μπορούμε δηλαδή να πούμε αν μας αρέσει ή όχι και να αρνηθούμε. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ενισχυμένη ευθύνη μεγαλύτερη ευθύνη. Αυτό σημαίνει ότι η μεγαλύτερη ευθύνη όμω φαίνεται να συνοδεύεται από, περισσότερη, από λιγότερη ενημέρωση. Για τις αλλιευτικές συμφωνίες πάντοτε ζητούσαμε πληροφορίε και αξιολόγηση, η οποία πάντοτε γινόταν από εξωτερικό συνεργάτη, ανεξάρτητο. Μιλάμε για εξωτερική ε, εταιρεία αξιολόγηση και τα απορίσματα αποστέλλονταν στο Ευρωκοινοβούλιο. Διεξοδικέ μελέτε, ε, εκατοντάδων σελίδων, με πολλέ πληροφορίε, πολλέ λεπτομέρειε. Μάλιστα ευχάριστε να τι διαβάζει κανεί και πολύ καλή πηγή πληροφοριών. Λοιπόν, από τότε που έχουμε την ε, διαδικασία τη σύμφωνη γνώμη, για κάποιο λόγο παίρνουμε μόνο μια περίληψη αυτών των μελετών, αυτών των εκθέσεων αξιολόγηση. Βλέπω λοιπόν με ιδιαίτερη χαρά που θέλει να μα ξεκουράσει, ότι θέλει να μα ξεκουράσει η Επιτροπή, όμω μα αφαιρεί τη δυνατότητα να διαβάσουμε και τι 200 σελίδε εφόσον το θέλουμε. Και το θέμα είναι ότι πρέπει να λάβουμε μια μορφωμένη απόφαση για το αν συμφωνούμε ή όχι με τις αλληλευτικές συμφωνίες. Αναρωτιέμαι λοιπόν, μπορεί να μα πει η Επιτροπή γιατί μα αποκρύπτει αυτέ τι αξιολογήσει. Είναι κάτι που απλώ τα μιλήσατε. Στο παρελθόν δεν φαίνεται να υπήρχαν τέτοια προβλήματα. Ξαφνικά τώρα που πρέπει να αποφασίσουμε φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν τη φιλοσοφία σας. Θα ήθελα λοιπόν η Επιτροπή να μας πει εάν θα μα στείλει και πάλι τι σχετικέ εκθέσει. Το λόγο έχει η Επιτροπή. Ο κύριος ε, Αλεξάνδρου, την ε, Κουσοπή. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Μια που παρουσιάσετε μια πολύ σωστή και ενδιαφέρουσα εισαγωγή για το πρωτόκολλο αυτό, επιτρέψτε μου εμένα να προσθέσω κάποιες πληροφορίες ώστε να γίνει περισσότερο κατανοητό το θέμα στα πλαίσια της Επιτροπής σας. Είναι αλήθεια ότι μιλάμε για αλλιευτική εταιρική συμφωνία. Είναι αλήθεια επίσης ότι διαπραγματευτήκαμε πέρυσι το Μάιο ένα νέο πρωτόκολλο τριετές. Εσείς και γραφήσατε τα κύρια σημεία της συμφωνίας αυτής. Οπότε εγώ απλώς θα σας πω ότι το συνολικό οικονομικό αντιστάθμισμα το ετήσιο εσείς αναφερθήκατε στο συνολικό ποσό για τρία χρόνια. Το ετήσιο αντιστάθμισμα είναι 615.250 ευρώ το χρόνο. Για να υπάρχει μεγαλύτερη ακρίβεια το λέω. Αυτό το οικονομικό αντιστάθμισμα και αυτή είναι η καινοτομία του πρωτοκόλου αυτού διαιρείται σε δύο τμήματα. Ένα τμήμα που είναι η πρόσβαση και ένα τμήμα που είναι η στήριξη του τομέα. Η προστιθέμενη αξία, αν θέλετε, το συν αυτού του πρωτοκόλου σε σχέση με το προηγούμενο είναι ότι επειδή έχουμε αυτή τη διάκριση, έχουμε εισαγάγει μία ρήτρα η οποία επιτρέπει ανα πάσα στιγμή να μπορούν οι υπηρεσίες της Επιτροπής να πάυσουν την πληρωμή του οικονομικού αντισταθμίσματος που προορίζεται για στήριξη του τομέα, εφόσον δεν καλύπτονται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια που έχουν συμφωνηθεί από κοινού ανάμεσα στην τρίτη χώρα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με άλλα λόγια δηλαδή, έχουμε στη διάθεσή μας ένα μέσο το οποίο δεν είχαμε κατά το παρελθόν για να πιέσουμε την τρίτη χώρα να τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε για στήριξη του τομέα. Στήριξη του τομέα που συνδέεται με την εθνική πολιτική για την Ελία ή με την εθνική στρατηγική της λόγω χώρας. Εννοείται ότι μιλάμε εδώ για ένα ποσό το οποίο μπορεί να φαίνεται μικρό σε σχέση με άλλες χώρες ή σε σχέση με άλλα επίπεδα πληρωμής. Όμως, μια που πρόκειται για στήριξη του τομέα, θα φροντίσουμε η δημοκρατία των Κομορών να διαθέσει σημαντικά ποσά, ακόμα και αν το σημαντικά είναι σχετικό, για την ανάπτυξη της αλίας και ιδιαίτερα για την ανάπτυξη της τοπικής αλίας, της μικρής κλίμακας αλίας. Θα ήταν πραγματι λυπηρό μέσα από τη συμφωνία αυτή να μην καταφέρουμε να συνεισφέρουμε έστω και σε ένα μικρό βαθμό στην ανάπτυξη της μικρής κλίμακας αλίας η οποία είναι αναγκαία για την περιοχή και όσον αφορά τις προτείνες που παίρνουν οι κάτοικοι και επειδή έτσι διαθέτουν έναν υπεύθυνο στόλο, έναν ε, στόλο στο αρχιπέλαγο των Κομορών. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας και τώρα θα απαντήσω στην ερώτηση του Ευρωβουλευτή για την έκθεσή ε, μας. Είναι αλήθεια ότι στείλαμε μια περίληψη. Περίληψη της ε, αξιολόγησης που ετοιμάστηκε από μια εξωτερική υπηρεσία. Ήταν μια περίληψη πράγματι. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα στείλουμε την ε, έκθεση ολόκληρη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εξάλλου, δεν είναι και το μόνο πρωτόκολλο για το οποίο έχουμε ετοιμάσει περίληψη. Εμείς περιμέναμε να έχουμε τα κύρια στοιχεία της διοργανικής συμφωνίας και γι' αυτό στείλαμε την περίληψη. Δεν ξεχάσαμε, δεν είναι επειδή δεν θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας τις πληροφορίες που έχουμε, στο κάτω-κάτω το έχουμε κάνει και κατά το παρελθόν. Απλώς θα σας στείλουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα ολόκληρη την έκθεση. Αυτά κυρία Πρόεδρε. Ελπίζω να ήμουν πλήρης. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Είναι σημαντικό να έχουμε αυτό το έγγραφο, πράγματι. Μπορώ να επιμείνω, κύριε εκπρόσωπε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να μας στείλετε όσο γίνεται πιο γρήγορα το έγγραφο αυτό. Σήμερα το βράδυ δυνατόν, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ή αύριο το πρωί το αργότερο. Γιατί έτσι, διαβάζοντά το, θα εμπνευστούμε να ετοιμάσουμε τι τροπολογίε μα. Βλέπετε και εμεί πιεζόμαστε από το χρόνο. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να έχω το περιεχόμενο τη έκθεση αυτή για να μπορέσουμε να είμαστε ενημερωμένοι και βάσει αυτή τη ενημέρωση να ετοιμάσουμε τι τροπολογίε μα. Εντάξει, μπορώ να βασιστώ σε αυτό που μα λέτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, θέλετε το λόγο. Α, παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, θα κάνω ό,τι μπορώ. Θα στείλω στις αρχές μου το έτοιμά σας όσο γίνεται πιο γρήγορα. Αυτό θα κάνω. Πρόεδρος, κοιτάξτε, δεν βλέπω γιατί το κοινοβούλιο που αποφασίζει με συναπόφαση για αυτό το θέμα πρέπει να δεχτεί περιορισμό στις πληροφορίες που παίρνει. Δεν βλέπω. Ειλικρινά ε, βασίζομαι ότι θα έχω την πλήρη έκθεση αύριο. Αυτό περιμένω. Κατά τα άλλα, σας υπενθυμίζω ότι πρέπει να ετοιμάσετε τροπολογίες και να τις υποβάλλετε πριν από την 7η Φεβρουαρίου. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα στις 3 Μαρτίου, ώστε να είμαστε έτοιμοι πριν αποφασίσει η Επιτροπή Αλίας. Ωραία, τελειώσαμε για σήμερα. Θα συνεχίσουμε αύριο το πρωί στις 9 με συνεδρίαση των συντονιστών. Και στη συνέχεια θα ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας στις 10.